Αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση. Σημείο 7 της ημερησίας διάταξης είναι η κατάσταση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων του τριμερούς διαλόγου. Κανονισμός κατά των βασανιστήριων μετά τον τρίτο τριμερή διάλογο την 1η Μαΐου, καταφέραμε να φτάσουμε σε πολιτική συμφωνία με το Συμβούλιο. Είναι ένα μεγάλο βήμα για τη βελτίωση των ελέγχων εξαγωγών ε, στα προϊόντα που είναι προϊόν βασανιστήριων και ε, θανατικής ποινής σε παγκόσμιο λοιπόν επίπεδο είναι ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω πως ήταν μεγάλη επιτυχία αυτή. Και η Μαρίτια Σάκε, η συγγήτρια, έχει συνεισφέρει σημαντικά σε αυτό. Συγχαρητήρια λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εντατική δουλειά που κάνατε. Θα θέλατε ίσως να προσθέσετε κάτι για αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα αρχίσω λέγοντας ότι ήταν ομαδική δουλειά. Ήταν μια προσπάθεια όλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα των σχεδόν εισηγητών και όλων όσοι εργάστηκαν σκληρά και ήταν κοντά στις διαπραγματεύσεις και στον τριμερή διάλογο. Είναι ένα από τα σπάνια χαρτοφυλάκια τα οποία έτυχαν μεγάλη πλειοψηφία εδώ στο Κοινοβούλιο. Πιστεύω πως ήταν μια πολύ καλή αφετηρία για τη διαπραγματευτική μας θέση με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Και τη χρειαστήκαμε και αυτό το μάθαμε πολύ σύντομα διότι ε, παρά την ε, απαγόρευση των αγαθών που προέρχονται από βασανιστήρια και από θανατική ποινή είναι κάτι που θεωρούμε δεδομένο, δεν ήταν τόσο εύκολη η εφαρμογή στην πράξη και οι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο. Ο πρώτος τριμερής διάλογος λοιπόν δεν είχε μεγάλη επιτυχία, ο δεύτερος ήταν εκρηκτικός θα έλεγα, αλλά μετά καταφέραμε να βρούμε ένα σημείο καμπής και το Συμβούλιο κατάλαβε τι χρειαζόταν. Ίσως πιέστηκε και από το χρονοδιάγραμμα και από το ότι σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να εξηγήσουν γιατί δεν επιθυμούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα. Επίσης, υπήρξε ανάγκη και για συμβιβασμούς. Αυτό σίγουρα δεν είναι το καλύτερο μέρος μιας διαπραγμάτευσης, όμως ένα σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι αναπόσπαστο κομμάτι της. Καταφέραμε λοιπόν ε, στο συμβιβασμό να συμπεριληφθούν ε, πολύ σημαντικά για το Κοινοβούλιο στοιχεία Καταφέραμε να δουλέψουμε πάνω σε πολύ βασικά θέματα. Ίσως να μην χρειαστεί να μπω σε λεπτομέρειες, ε, κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω για όσους δεν ήταν εκεί. Καλύτερα θα ήταν να σταματήσω εδώ, να ολοκληρώσω λέγοντας ότι καταφέραμε να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα όπου οι παγκόσμιες αξίες, τα παγκόσμια ανθρώπινα δικαιώματα σε σύνδεση με τους ε, κανόνες του εμπορίου ε, κατάφεραν να βελτιωθούν. Ελπίζω λοιπόν να το καταλάβουν όλοι αυτό και να κάνει τη διαφορά και σε άλλα μέρη του κόσμου όπου οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν τη θανατική ποινή βασαριστήρια. Ελπίζω λοιπόν να γίνει ε, αισθητή η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ Μαρίτια. Πράγματι θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν σχόλια από τους Κιώδης. και εγώ να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί νομίζω ότι θα θαυμάσια η εργασία της και υπερασπίστηκε τη θέση του Κοινοβουλίου και όπως μας εξήγησε δεν ήταν εύκολο. Επιπλέον η στάση της ήταν ε, θετική για ανοιχτό διάλογο με όλες τις πολιτικές ομάδες έτσι μπορέσαμε να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε ως ομάδα πολύ επικοδομητική και ευχάριστη αυτή και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον πρόεδρο Λάνια που νομίζω ότι έκανε πολύ σημαντική εργασία και ιδιαίτερα για να υπερασπιστούμε τις εξουσίες του Κοινοβουλίου, την δυνατότητα να συμμετάσχουμε στην ομάδα συντονισμού, για την παρακολούθηση εφαρμογή του νέου κανονισμού και επίσης ε, όλες τις ε, μη κάπα που συμμετείχαν και ιδιαίτερα την εργασία που κάνει η Διεθνής Αμνηστία και το Ίδρυμα ΟΜΕΓΑ. Όπως είπε και η συγγήτρια, πρέπει να θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό το μεγάλο βήμα προόδου για την Ένωση. Επειδή ορισμένοι υποτιμούν την Ευρώπη και προσπαθούν να μειώσουν ε, την αξία της, είναι, τις αξίες της μάλλον, είναι σημαντικό νομίζω να δείξουμε ότι τις πειρασπιζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να αδιαφορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για βασανισμούς και θανατικές ποινές και έτσι δεσμευόμεθα να ε, ελέγχουμε το εμπόριο των ε, εργαλείων, των μηχανισμών, των προϊόντων που ε, χρησιμοποιούνται για βασανιστήρια και εκτελέσεις θανατικής ποινής και νομίζω ότι στόχος μας πρέπει να είναι να επιτύχουμε σχεδόν πανψηφία για το κείμενο αυτό και θα άξιζε τον κόπο. Ευχαριστώ κύριο Φίσας. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την συγκήτρια για την εργασία της. Ήταν ε, ευχαρίστηση να συνεργαστούμε μαζί της για αυτό το σημαντικό θέμα και με τους άλλους κοιόδης φυσικά. Νομίζω ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια, όπως είπε σωστά και η συγκήτρια, η επίτευξη της ενότητας μαζί με την στήριξη του Προέδρου. Όλα αυτά ήταν αποφασιστικά, ούτω ώστε να πιστεί και η Κομισιόν μετά από πίεση για να δεχθεί τη θέση της Επιτροπής μας του Κοινοβουλίου. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και μερικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Εγώ εργάστηκα με την ε, Βρετανική ΜΚΟ Retrieve, η οποία επίσης ε, ήταν ιδιαίτερα μετριοπαθής, ε, δεν είχε ακραίες θέσεις και είναι σημαντικό τόνισε και εκείνη και μας βοήθησε για να εμποδίσουμε το εμπόριο σε αυτούς τους μηχανισμούς. Και θα πρέπει να αποκαλέ, αποτελέσει προηγούμενο αυτή η συμφωνία και για άλλες συμφωνίες για θέματα διεθνούς εμπορίου και πρέπει να επαγρυπνούμε όταν υπογράφουμε συμφωνίες με χώρες οι οποίες εφαρμόζουν βασανισμούς, ακόμη και νομοτύπος για ορισμένες ποινές. Είναι σημαντικό λοιπόν αυτό και επαναλαμβάνω πρέπει να επαγρυπνούμε να έχουμε τις αναγκαίες ρήτρες διαφύλαξης στις συμφωνίες διεθνούς εμπορίου με τις χώρες που δεν σέβονται ε, κατά ελάχιστον τα ανθρώπινα δικαιώματα στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τα επόμενα βήματα λοιπόν είναι έγκριση από το Συμβούλιο, από την Κορεπέρ στις 13 Ιουνίου, 30 Ιουνίου και μετά θα περάσουμε στις διαπραγματεύσεις τριμερούς διαλόγου. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 14 Ιουλίου. Και μετά μπορούμε να πάμε στην Ολομέλεια. Πολύ ωραία. Επόμενος συνεχίζομενος τριμερής διάλογος για τα ορυκτά που αποτελούν ε, αντικείμενο σειράξεων. 11 Μαΐου έλαβε χώρα και είχαμε δείξει πνεύμα συνεργασίας, συμβιβαστικό πνεύμα, φτάσαμε πολύ κοντά σε έναν συμβιβασμό στα κεντρικά σημεία, αλλά όχι τόσο κοντά ώστε να συμφωνήσουμε στα πάντα. Και Σήμερα το βράδυ θα διεξαχθεί ένας άλλος τριμερής διάλογος, θα είναι μια τελευταία προσπάθεια. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη σχετική ε, διαπραγμάτευση. Αλλά θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πραγματικά ε, χαίρομαι κι εγώ και συμμερίζομαι την αισιοδοξία σας ε, όταν λέτε ότι θα είναι ο τελευταίο τριμερής διάλογος, όντω θα είναι ο τελευταίος, ε, θα υπάρξει συμφωνία και βέβαια μετά θα υπάρξει πολύ τεχνική εργασία που θα πρέπει να γίνει επί του κειμένου και ούτω καθεξής. Άρα θα περάσουμε κατά πάσα πιθανότητα στη Σλοβακική ε, Προεδρία, όμως το βασικό πλαίσιο της συμφωνίας νομίζω ότι θα μπορέσει να θεσπιστεί σήμερα το απόγευμα. Ίσως ε, να πρέπει να σας μιλήσω για κάποια βασικά στοιχεία σύντομα της, ε, του συμβιβασμού, μάλλον όχι του συμβιβασμού, της συμφωνίας που θα γίνει σήμερα το βράδυ. Καταρχάς, όλοι οι κανονισμοί θα πρέπει ως ε, βασικό του στοιχείο να έχουν τη συμμόρφωση με τις κατευθυντές γραμμές του ΑΣΑ. Επίσης, διάφορα προγράμματα δέουσας επιμέλειας που θα πρέπει να είναι βασικά στοιχεία των κανονισμών επίσης, η ιδέα της του υποχρεωτικού δικαστικού ελέγχου και για το ε, κομμάτι της αλυσίδας εφοδιασμού πριν ε, από την ε, πώληση. Αυτά όλα πρέπει να γίνουν βάση λοιπόν της δέουσας επιμέλειας και του νομικού ελέγχου. Υπάρχουν ε, επίσης κάποια τεχνικά στοιχεία ε, για τις ε, μεθόδους ανάθεσης, για τα αποθέματα που δίνουν πολύ ξεκάθαρη ένδειξη για το τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει να γίνεται ε, Ω προ την προστασία και εκτιμένων δικαιωμάτων και Και επίσης έχουμε και μια πολύ σημαντική ρήτρα αναθεώρησης που είναι πολύ σημαντικό στοιχείο γιατί ε, μερικά χρόνια ε, μετά την έναρξη ισχύω του κανονισμού θα μπορούμε να δούμε τις επιπτώσεις επιτόπου και στη βιομηχανία. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία νομίζω. Ε, αυτή η συμφωνία ελπίζω ότι θα ολοκληρωθεί όπως είπα σήμερα το βράδυ και θα αποτελέσει τη βάση ε, για να έχουμε έναν ε, αποτελεσματικό κανονισμό με τον οποίο θα μπορούμε να δουλέψουμε. Ευχαριστούμε. Ο Μάικ. Η Μάικ. Ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο, διότι ε, αυτό το θέμα ήταν πολύ πιο δύσκολο από τα προηγούμενα. νομίζω, απλώς να το ελέγξω λίγο και με τον εισηγητή, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του περιεχομένου, ε, το οποίο τώρα λέτε ότι θα ψηφιστεί ε, συμπίπτει με αυτά που είχαμε στην Επιτροπή ΙΝΤΑ ήδη ψηφίσει. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη ερώτηση ίσως να μην έχει τόσο νόημα γιατί αυτοί που έχουν τις πιο ισχυρές απόψεις δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή για να σκεφτούν. Ίσως όμως πρέπει κάποια στιγμή να σκεφτούμε πώς ψήφος μας στο Κοινοβούλιο εδώ μας ε, ισχυροποιεί από αποδυναμώνει τη θέση μας ε, στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Να πάρουμε τα μαθήματα που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε στο μέλλον. Ε, να απαντήσουμε άμεσα. Ε, ναι. Ε, ως προς τα αποτελέσματα στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, όχι, εργαζόμαστε επί ενός πιο ισχυρού κειμένου δεν είναι αυτό ακριβώς που ψηφίσαμε. Ε, όχι, ε, γιατί εμείς ψηφίσαμε την πλήρως εθελούσια προσέγγιση που προτάθηκε στο Ινολομέλεια του Κοινοβουλίου, αλλά τώρα είναι μια διαδικασία η οποία είναι υποχρεωτική για τις εταιρείες ε, που είναι στην αλυσία εδα αξίας, στην πάνω πλευρά δηλαδή, από την εξόριξη και μετά. Ε, υπήρξαν πολλές αλλαγές ε, στο διάλογο. Ε, Φτάνουμε μέχρι το χιτήριο. Υπήρχαν πολλές αλλαγές λοιπόν στο διάλογο που είχαμε στην Επιτροπή μας. Είχαμε να κάνουμε με τα προγράμματα της δέουσας επιμέλειας εκεί που θα πρέπει να εφαρμόζει βιομηχανία και αυτό τελικά στο μεταξύ έγινε το κεντρικό στοιχείο των συζητήσεων στον τριμερή διάλογο. Επίσης, νομίζω ότι ε, δόθηκε προσοχή στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, να μην υπάρχει ε, υπερβάλλον υπερβάλλουσα γραφειοκρατία. Ε, όλα αυτά ε, άλλαξαν σε σχέση με το παράρτημα του κανονισμού. Ε, δεν είναι ακριβώς το ίδιο κατόφλι για τα διάφορα προϊόντα φυσικά, δεν μπορεί να είναι το ίδιο, αλλά θα είναι ένα κατόφλι το οποίο θα καλύπτει τη μεγάλη πλειοψηφία, το 95 περίπου των εισαγωγών αλλά οι μικρές επιχειρήσεις δεν θα επιβαράνονται με την, με γραφειοκρατία. Για την ψήφο μας τώρα στο Κοινοβούλιο. Μόλις, δίνουμε, μόλις δούμε τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα, θα μπορώ να σας απαντήσω. Αν επιτύχουμε, σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο τα πήγε καλά. Είχαμε στην αρχή μεγάλες προσδοκίες και μετά δείξαμε ευελιξία. Να σας πω όμως την αλήθεια, αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα κάποια απόσταση μεταξύ των κρατών μελών της Προεδρίας ε, του Κοινοβουλίου φυσικά και των αρχικών προσδοκιών του Κοινοβουλίου. Εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δείχνουμε ευελιξία μεν, από την άλλη τα κράτη-μέλη πρέπει να αυξάνουν το επίπεδο αποδοχής ε, της ευθύνης ε, ως προς τον κανονισμό. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρίγκλερ. Για να δούμε τι θα γίνει απόψε. Ωραία. Πάμε τώρα στο σημείο 8. Αντιπροσωπεία ad hoc στη Σεούλ, Δημοκρατία της Νοτιού Κορέας, 17 με 19 Μαΐου. Ήμουν ε, επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας. Είχα αυτή την τιμή, ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη. Ο σκοπός της αντιπροσωπείας ήταν να δει ακριβώ ε, ποια είναι η εμπειρία από τη Συμφωνία Εμπορίου με την Νότια Κορέα που ισχύει εδώ και πέντε χρόνια. Ε, συζητήσαμε επίσης κάποιες βελτιώσεις περαιτέρω και εξελίξεις αυτής της συμφωνίας. Είχαμε μια αντιπροσωπεία με όλα τα κόμματα και όλες τις εθνικότητες. Είχαμε επίσης και τον ε, πρόεδρο της, Επιτρο... της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κορέα και συναντηθήκαμε με υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, τον ε, Υπουργό Γεωργίας για παράδειγμα, ε, Συζητήσαμε την πολιτική γεωργίας, τις πατάτες, Είχαμε επίσης ε, μέλη ε, της ε, βιομηχανίας, εμπορίου, της του εμπορικού κόσμου, είχαμε εισαγωγείς, είχαμε προσώπους από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, επίσης μέλη των εγχώριων συμβουλευτικών ομάδων, επίσης τον πρέσβη των ΙΠΑ διότι σχετίζεται η Νότιος Κορέα με τις εξελίξεις στις Ηνωμένε Πολιτείε και επίσης ε, συζητήσαμε γενικότερα τις σχέσεις, τις εμπορικές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νοτιού Κορέας. Ήταν πολύ επικοδομητική συζήτηση. Ε, μας έδωσε μια πλήρη εικόνα. Επίσης επισκεφθήκαμε μια βιομηχανική ζώνη που έκλεισε από τον Φεβρουάρι. Θέλαμε να πάμε εκεί, αλλά μπορέσαμε μόνο να δούμε λίγο ε, το κομμάτι στην αποστρατικοποιημένη ζώνη. Μου θύμισε λίγο την κατάσταση ε, που είχαμε στην Γερμανία με πριν το 1989 με τα δύο γερμανικά κράτη. Είχα την εντύπωση ότι δεν υπήρχε σωστή παρακολούθηση της διαδικασίας ε, εφαρμογής. Ε, τα εργασιακά δικαιώματα επίσης είναι προβληματικά. Άρα, ως προς την βελτίωση της συμφωνίας, η κορεάτικη πλευρά μας είπε ξεκάθαρα ότι θα θέλει ένα κομμάτι επενδυτικό στη συμφωνία που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και από την άλλη ε, υπήρξαν κάποια λιγότερο σημαντικά στοιχεία. Για παράδειγμα, ε, η ρήτρα ε, για τις άμεσες μεταφορές, δηλαδή μόνο τα προϊόντα που έρχονται από την Κορέα απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτονται και τα τούμπαλιν. ένα άλλο προϊόν ας πούμε που θα πήγαινε από τη Σιγκαπούρη στην Νότια Κορέα, ίσως θα πρέπει και αυτό να καλύπτεται. Επίσης, ε, επισκευές προϊόντων και μηχανημάτων θα πρέπει και αυτές να καλύπτονται. Έγινε μια γραπτή έκθεση, αλλά έχουμε τον εισηγητή μας εδώ, ο οποίος θα μπορούσε να κάνει κάποια επιπλέον σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτήν την επίσκεψη που ήταν πολύ καλά οργανωμένη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν τον Πρόεδρό μας που ε, ηγήθηκε με θαυμάσιο τρόπο αυτής της ε, αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ τη γραμματεία μας, τους συμβούλους μας, ε, όλο το προσωπικό που βοήθησε. Η επίσκεψη αυτή, όπως είπα, ήταν πολύ καλά προπαρασκευασμένη, όχι μόνο από πλευράς λεπτομεριών διεξαγωγής, αλλά και όσον αφορά το πρόγραμμα. Όλα ήταν πολύ σωστά προετοιμασμένα οι συνομιλητές μας είχαν επιλεγεί πολύ σωστά. Όλα αυτά καταδεικνύουν ότι τέτοιες επισκέψεις πρέπει πάντα να είναι καλά προπαρασκευασμένες. Ήδη ε, από τις Βρυξέλλες, πριν ξεκινήσουμε να τις προετοιμάζουμε. Πριν ξεκινήσουμε, οπωσδήποτε. Ε, γιατί οι αποφάσει που έπρεπε στι Βρυξέλλε μετά έχουν επίπτωση στο, στο τι συμβαίνει επί τόπου. Για την ε, Συμφωνία Ελευθερών Μπορείου με εξέπληξε ότι η στάση που εξέφρασαν οι συνομιλητές μας επί τόπου δεν είναι η ίδια με τη στάση τους στις Βρυξέλλες. Εδώ είναι πιο άκαμπτη, πιο ακραία ορισμένες φορές η στάση τους και ε, πολύ συχνά είναι επικριτική. Έτσι φέρονται στις Βρυξέλλες. Αλλά όταν πας εκεί, στη Νότια Κορέα, διαπιστώνεις ότι είναι διαφορετική η στάση τους. Ε, είναι σαφές ότι είναι πολύ ικανοποιημένοι οι εταίροι μας από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για αυτήν την συμφωνία. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πολύ μεγάλη ε, απόκληση μεταξύ τη στάση τους εδώ και εκεί. Επίσης είναι ενδιαφέρον ότι είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με όλους όσους συμμετέχουν, όλους όσοι συμμετέχουν στην ε, εφαρμογή της ε, Συμφωνίας Ελευθερών Μπορείου. Συναντηθήκαμε με τους αρμόδιους υπουργούς, ε, βιομηχανίας, εμπορίου, γεωργίας, εξωτερικών, όλους τους εταίρους όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία. Επίση είδαμε εκπροσώπους ε, της βιομηχανίας. Και επίσης συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους ε, των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ε, δραστηριοποιούνται στη Νότια Κορέα. Εάν λοιπόν περιοριζόμασταν ε, να επιχειρούμε να συνοηθούμε με τους εταίρους μας αυτούς ε, μόνο στις Βρυξέλλες, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα ε, που είχαμε να κάνουμε τις επαφές εκεί με τα συνδικάτα, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Είναι δύσκολο να έρθουν όλοι αυτοί στις Βρυξέλλες. Ενώ, χάρη στη δική μας επίσκεψη, τους είδαμε τη θέμενη αξία. Γιατί αυτά που μας είπαν πρέπει οπωσδήποτε να παίξουν το ρόλο τους στη σχέση μας με την Νότια Κορέα. Δηλαδή τις ενδεχόμενες προσαρμογές ε, ε, για διάφορα θέματα εργασιακού δικαίου, εργασιακών δικαιωμάτων κτλ. Ε, πρέπει να σας πω ειλικρινά ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συμφωνία αυτή στην οποία καταλήξαμε και από το πώς εφαρμόζεται. Δεν είναι μόνο θέμα στατιστικών στοιχείων. Πρέπει να μπορεί να ερμηνεύει σωστά τα στατιστικά στοιχεία Πρέπει να έχεις ε, την κατάλληλη πείρα για να δεις ε, την ε, θετική επίπτωση αμοιβαία εποφελών σχέσεων και πρέπει να μπορείς να δεις αν αυτές οι θετικές εξελίξεις σχετίζονται με τη Συμφωνία Ελευθερομπορίου ή είναι απλώς μια γενική τάση που έχει να κάνει με τη γενικότερη συγκυρία στις αγορές. Αλλά πέρα από αυτό, τονίζω ότι τα μακροοικονομικά στοιχεία είναι πολύ ενθαρρυντικά. Έχοντας μιλήσει λοιπόν με όλους τους ενδιαφερομένους, πρέπει να πω ότι είναι γενικότερα ενθαρρυντική, ενθαρρυντική η κατάσταση εκατέρωθεν. Νομίζω ότι και εκατέρωθεν μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι από αυτά που επιτύχαμε. Αλλά φυσικά έχουμε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους. Για παράδειγμα, για τα εργασιακά δικαιώματα, την ενίσχυση της δημοκρατίας, της κοινωνίας των πολιτών από τη μία και από την άλλη περισσότερο ε, δίκαιους κανόνες θεμητού ανταγωνισμού. Αυτές είναι πλευρές που πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω. Είπαμε, τα δικαιώματα των εργαζομένων, οπωσδήποτε, και η δυνατότητα παρέμβασης της κοινωνίας των πολιτών. Εδώ απέχουμε ακόμη πολύ από μια άρεστη κατάσταση. Και για τις προσδοκίες ε, των δύο συμβαλωμένων θέλω να πω ότι οι Κορεάτες συνομιλητές μας συχνά μας ανέφεραν ότι θα έπρεπε να γίνουν προσαρμογές στη συμφωνία για να προστατευτούν οι επενδύσεις. Αυτό πρέπει να τεθεί, αλλά δεν είναι εύκολο θέμα. Αντίθετα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Σε αυτή τη φάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε σε φάση επανακαθορισμού των θεμάτων προστασίας των επενδύσεων και των μηχανισμών επίλυσης διαφορών επ' αυτών. Και επίσης ε, για πολλά κοινωνικά θέματα ε, πρέπει να ξαναδούμε. Λοιπόν, θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Να σας πω τι πρόκειται να κάνουμε τους επόμενους μήνες, στο εγγύ μέλλον δηλαδή. Ο πρόεδρος ε, και άλλοι συνάδελφοι, αν έχετε προτάσεις, παρακαλώ να ε, με ενημερώσετε. Τον Ιούλιο, 13-14, θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή μας και κατόπιν τον Οκτώβριο 12 και 13 θα συζητήσουμε την έκθεση θα υποβληθεί, θα εξεταστεί κατόπιν θα ψηφίσουμε κατά τη συνεδρίασή μας στις 28-29 Νοεμβρίου και τέλος, τέλος την Ολομέλεια κατά την ε, εβδομάδα 12 με 15 Δεκεμβρίου. Και αν δεν ε, προλάβουμε τον Ιανουάριο του 17. Α, αυτά είναι τα σχέδια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Σένφελ για αυτήν την παρουσίαση της δουλειά που έχει γίνει ε, εν ώψη της έκθεσης την εμπορική συμφωνία. Υπάρχουν άλλα σχόλια. Ο κύριος Σούστερ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο θέματα τα οποία ήδη έχουν ε, αναφερθεί, αλλά θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντικά για μένα. Εργασιακά δικαιώματα. Πιστεύω ότι στο παρελθόν ε, δεν έχουμε δώσει τη δέουσα προσοχή και πρέπει να το κάνουμε αυτό τώρα. Ε, σίγουρα πρέπει να τηρούνται οι κανόνες του ΠΟΕ αλλά πρέπει να επανεξετάσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν περιπτώσεις μέλων, ε, συνδικαλιστικών οργανώσεων που έχουν συλληφθεί ε, λόγω της δραστηριότητάς τους. Ε, όταν αυτό λοιπόν είναι ε, λόγος σύλληψης, το να ανήκει δηλαδή κάποιος ε, σε συνδικαλιστική οργάνωση και να καταλήξει στη φυλακή, τότε βλέπουμε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και πόσο ε, επίκουσα είναι η ανάγκη να συζητηθούν. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, πρέπει μάλλον να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση για να καταστεί αυτό σαφές. Έπειτα θα ήθελα να σταθώ στην προστασία πενδύσεων. Πιστεύω πως ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι κορεάτε θεώρησαν αυτό ως αφετηρία των συνομιλιών, ότι θέλουν προστασία για τις επενδύσεις τους, προστασία των επενδυτών, αλλά από την άλλη μου φαίνεται ότι στην παλιά συμφωνία υπάρχουν τέτοια στοιχεία τα οποία στηρίζονται ε, στα οποία στηρίζονται και είναι κάπως ε, παράλογα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω πως αυτό μου φαίνεται λυπηρό και μου φαίνεται επίσης δυσάρεστο ότι οι Κορεάτες δεν έχουν φτιάξει κάποια, κάποιο νέο δικαστικό μηχανισμό για ε, αυτή την προστασία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως θα έπρεπε να συζητηθεί. Ευχαριστώ πολύ. Αν θυμάμαι καλά, η Κορέα έχει 22 εμπορικές συμφωνίες με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι αρκετά δύσκολο έργο να βελτιωθεί το σύστημα. Ο κύριος Μπούχνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Νομίζω πως όλα λίγο πολύ έχουν υποθεί. Βρίσκω αρκετά ευχάριστο ότι με αφορμή το εμπόριο, την εμπορική συμφωνία, μπορούμε να αποκομίσουμε ε, πολύ θετικά ε, στοιχεία. Η κατάσταση με τα εργασιακά δικαιώματα στην Κορέα είναι κάτι που έχει ήδη αναφερθεί. Τα εργασιακά δικαιώματα καθ' αυτά στην Κορέα δεν ε, αντιστοιχούν με τα δικά μας πρότυπα. Δεν είναι στα ίδια επίπεδα με τα δικά μας. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, υπάρχουν εργαζόμενοι, κάτι σαν τους γκασταρμπάιτερ, εποχιακοί εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται σε συνθήκες σχεδόν ε, δουλείας. Είναι, ε, τους πληρώνουν τα εισιτήρια για να φτάσουν στην Κορέα. Ο μισθός είναι εξαιρετικά χαμηλός. Μόλις φτάνουν στη χώρα τους παίρνουν τα διαβατήρια. Δεν μπορούν ε, να αλλάξουν εργοδότη αυτοί οι άνθρωποι εάν το επιθυμούν. Ε, πέφτουν θύματα στιγμής εκμετάλλευσης, ιδιαίτερα στην γεωργία. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνουν ψεκασμούς χωρίς καμία απολύτως προστασία. Δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καμία ασφάλεια, καμία προστασία. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για μας, διότι η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου αφορά ακριβώς προϊόντα τα οποία έχουν ε, παραχθεί με τέτοιον τρόπο. Εδώ δηλαδή νομίζω πως ε, πρέπει η Ευρώπη να κάνει κάτι εάν θέλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα πρότυπα τα οποία, ε, για τα οποία είμαστε τόσο περήφανοι. Ευχαριστώ. Ωραία. Ολοκληρώνω λοιπόν αυτό το σημείο μετά από αυτήν την παρέμβαση και περνάω στο σημείο 9. Η αποστολή αντιχώ hoc στην 11η συνεδρίαση τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΠΟΑΣ, 13 και 14 Ιουνίου στην Γενέβη. Δευτέρα και Τρίτη δηλαδή, αυτή τη εβδομάδα. Νομίζω πως η συνέλευση αυτή τη φορά ήταν πιο ζωντανή από τα προηγούμενα έτη. Είχαμε δείγματα πιο ενεργού δράσης από, τα άλλα, από τους άλλους συμμετέχοντες, από τα άλλα κράτη. Υπήρχαν προετοιμασμένες δηλώσεις από τις ε, κυβερνήσεις τους μέχρι πρότινος. Τώρα όμως είδαμε να έχει αλλάξει αυτό. Είδαμε πρωτοβουλία και με χαρά μου το διαπίστωσα. Συζήτησα με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΠΟΕ για το μέλλον του ΠΟΕ. Υπήρχαν παρεμβάσεις από βουλευτές, από εμάς, ο κύριος Ρούμπιγκ και ο κύριος Σόλτς μας εκπροσώπησαν και στις παρεμβάσεις μας σταθήκαμε στους ε, στόχους πέρα από τον Αϊρόμπι. Νομίζω πως ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα. Νομίζω σας έχει διανεμηθεί κιόλα. Το Κοινοβούλιο λοιπόν έπαιρξε ενεργό ρόλο στις συζητήσεις για την στρατηγική μετά το Ναϊρόμπι. Επίσης κατέστησε σαφές ότι χρειάζονται μεταρρυθμίσεις και χρειάζεται επίσης να δούμε με μεγαλύτερη προσοχή τις ε, διμερείς σχέσεις στα πλαίσια του ΠΟΕ. Είμαι αρκετά ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα λοιπόν του συνεδρίου και αυτό επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της κοινοβουλευτικής συνέλευσης, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία του ΠΟΕ, υπήρξε ξεχωριστό φόρουμ αφιερωμένο στο φύλλο και το εμπόριο. Και συνάδελφος Ροντρίγκε μάλιστα ασχολήθηκε με αυτό. Και με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα ότι συνάδελφοι από την Τινησία, από την Ινδονησία, από διεθνείς οργανισμούς ήταν εκεί και εστίασαν στη διάσταση του φύλου στα πλαίσια των εμπορικών διαπραγματεύσεων. Ήταν λοιπόν μεγάλη μου χαρά που κατάφερα να ακούσω αυτές τις ε, συζητήσεις, αυτές τις απόψεις και αυτό νομίζω διαφαίνεται και στο τελικό κείμενο. Ήταν, όπως σας είπα, μία ενημέρωση για την ad hoc ε, αποστολή. Θα λάβετε γραπτό κείμενο, αλλά δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιο μέλος της αποστολής να προσθέσει κάτι, ο κύριος Ρούμπικ. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω διότι αυτή η αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ε, απέδειξε ότι μπορεί να συνεργαστεί πολύ καλά με τα υπόλοιπα μέλη της ε, συνέλευσης. Έχουμε δει ότι αυξάνεται το ενδιαφέρον για το μέλλον του εμπορίου και αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη δημιουργία ενός σωστού ε, θεσμικού πλαισίου. τώρα, συζητήθηκε πολύ έντονα το θέμα του Brexit και πώς αυτό θα ε, επηρεάσει τις λειτουργίες του ΠΟΕ, ποιο μοντέλο σε περίπτωση Brexit θα επιλέξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά συζητήθηκε πολύ το θέμα της προσφυγικής κρίσης και αυτό μέσω της διάστασης του ΠΟΕ. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι συνομιλίες. Ωραία. Κάποιος άλλος? Εκτός μικροφώνου, Πρόεδρος. Πάμε τότε στο σημείο 10. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας, η οποία έχει να κάνει με τις αλλαγές, την τροποποίηση των ε, παραχωρήσεων που προβλέπονται στον πίνακα τη Δημοκρατία τη Κροατία, στο πλαίσιο τη προσχώρηση τη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Ρίγκλερ είναι ο εισηγητή. Θα του δώσουμε το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ, συνάδελφοι. Με την προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε η Δασμολογική Ένωση. Σύμφωνα με τους κανόνες ε, του ΠΟΕ θα έπρεπε να γίνουν κάποιες ε, διαπραγματεύσεις για το δασμολογικό πίνακα για την έτσι, Κροατία έτσι ώστε να έχουμε μια αντισταθμιστική προσαρμογή που πρέπει να υπάρξει κάθε φορά ε, που υπάρχουν περισσότεροι δασμοί για την χώρα που προσχωρεί πέρα από τα επίπεδα που ήταν ήδη συμφωνημένα στα πλαίσια του ΠΟΕ. Τον Ιούλιο του 2013 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις ε, και ως αποτέλεσμα αυτών η Επιτροπή πρότισε στο Συμβούλιο να υπογράψει μια συμφωνία υπό τη μορφή ανταλλαγής επιστολών που θα γινόταν παράλληλα με μια άλλη πρόταση που κατατέθηκε στο Συμβούλιο και εγκρίθηκε με την ε, σύναψη αυτής της συμφωνίας. Τα αποτελέσματα της συμφωνίας θα έπρεπε να ε, γίνουν ε, ως εξής ε, να έχουμε κάποιους δασμούς για τα υποδήματα, για τις ε, συσκευές κλιματισμού. Επίσης στις γεωργικές ποσοστώσεις θα υπήρξε μια αύξηση που θα έπρεπε η Επιτροπή να συμπεριλάβει σε ένα νέο εκτελεστικό κανονισμό, κάποιες αλλαγές σχετικά με το σκόρδο και τα μανιτάρια επιπλέον. Σύμφωνα με το άρθρο 14 ε, της ε, Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου, η ε, Κίνα είχε το δικαίωμα αποκατάστασης των προηγούμενων δικαιωμάτων της και γι' αυτό εμείς και εγώ συγκεκριμένα προτείναμε να γίνει αυτή η αλλαγή βάσει της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου. Επίση, η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων έχει κάνει γνωμοδότηση που είναι θετική. Οπότε συστήνω στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια στη συνέχεια ε, να δοθεί η συνένεση ε, του Κοινοβουλίου. Ε, και με αυτό το πνεύμα έχω συντάξει και τη σύστασή μου. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στους Σκιώδης. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ε, είναι πολύ συγκεκριμένα τα σχόλια ε, που έχουν ακουστεί, οπότε απλώς θα ήθελα να υποστηρίξω τη σύναψη της συμφωνίας, η ΕΜΑ. Το ίδιο και για το ECR, υποστηρίζουμε τον εισηγητή και μπορούμε να δώσουμε τη συνένεσή μας στο Κοινοβούλιο, νομίζω. Ευχαριστώ, κύριος Λάμπς δεν είναι εδώ, κύριος Σόλτς, ο κύριος Μπούχνερ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα συνενέσουμε. Και δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να έχει ζητήσει το λόγο, οπότε δίνω το λόγο στην Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα απλώς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εργασία του επί αυτού του θέματος και αναφέρω, να αναφέρω ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα ε, την όλη διαδικασία που ακολουθεί τη προσχώρηση τη Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φαντάζομαι ότι όλε οι διαδικασίε θα γίνουν ομαλά. Στο εξή. ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόκ από την Επιτροπή ΑΦΕΤ μου έστειλε επιστολή και μου λέει ότι με μεγάλη του χαρά θα συνενέσει και αυτός στη συμφωνία. Κύριε Βίγκλερ, θέλετε να πείτε κάτι έτσι ως κατάληξη. Όχι, απλώς να ευχαριστήσω για την υποστήριξη των σκιωδών. Ευχαριστώ. Η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες είναι Παρασκευή 17 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα. Σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Το μέλλον των σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020, μετά την ε, συμφωνία του Κοτονού, ε, που θα, μετά την εκνοή μάλλον της συμφωνίας του Κοτονού. Η ΔΕΒΕ κάνει μία έκθεση για αυτό το θέμα πρωτοβουλίας και έχουμε ε, ως ε, εισηγητή τον Πέντρο Σίλβα Περέα για αυτό το θέμα. Ε, δεν είναι εδώ, αλλά ο Ντέβιτ Μάρτιν θα τον αντικαταστήσει. Ναι, μάλλον ο Πέντρο είναι στο Windhoek τώρα, ακριβώς στη συνάντηση της κοινής, ε, της μικτής κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Θα σας διαβάσω τη δήλωσή του λέει ότι η συμφωνία αυτή είναι μια αξιόλογη συμφωνία, βιώσιμη, πρέπει να την στηρίξουμε και τονίζει ότι το εμπόριο είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της διαδικασίας κοτονού και αυτή η διάσταση θα πρέπει να είναι τμήμα ή ε, ασδήποτε Συμφωνία συμφωνίες 31 Μαΐου είχε τη δυνατότητα να κάνει μια άτυπη ανταλλαγή απόψεων με τι πολιτικέ ομάδε για το σχέδιο γνωμοδότηση, που ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η συνάντηση και συνεχίζει τη συζήτηση με βάση τα αποτελέσματα αυτής της διαβούλευσης. Η σχέση με τις χώρες ΑΚΕ ξεκίνησε το 1975 και από το 2000 αυτή η συνεργασία διοικείται από τις εταιρικές συμφωνίες Κοτονού που όπως είπατε εκπνέει στις 29 Φεβρουαρίου 2020. Αυτό το μήνα περιμένουμε μια αξιολόγηση της συμφωνίας που θα εκτιμήσει, σε τι, έχει επιτύχει, αν έχει επιτύχει τους στόχους της, θα κάνει απολογισμό των διδαγμάτων και θα μας δώσει διδάγματα για το μέλλον. Αυτή η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική φάση για την μετακοτονού περίοδο. Πριν μιλήσουμε για θέματα εμπορίου, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις απόψεις του χρόνων και για το μελλοντικό πλαίσιο. Η βασική συζήτηση της, κοινής, της μικτής κοινοβουλευτικής συνέλευσης που λύγει σήμερα είναι ακριβώς το μέλλον αυτής της σχέσης μετά τη λήξη της Συμφωνίας Κοτονού και είναι κατάλληλη στιγμή γιατί έγινε η συνάντηση κορυφής των χρόνων ΑΚΕ στην Παπουασία Νέα Γουινέα που μια ομάδα διακεκριμένων προσωπικότητων έκανε μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό Όσον αφορά το εμπόριο και τις οικονομικές πλευρές, τονίζει ότι η Ένωση είναι από τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους και πρέπει να καταλάβουμε ότι η βιομηχάνηση και η διαφοροποίηση των οικονομιών τους, των χωρών ΑΚΕ, είναι ακόμη περιορισμένη και το εμπόριο πρώτων υλών είναι ένα μεγάλο τμήμα του εμπορίου των χωρών ΑΚΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το καθεστώ εμπορίου αναθεωρήθηκε για να είναι συμβατό με του κανόνε του ΠΟΕ και οι εξαγωγέ των χωρών αυτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπόκεινται σε διαφορετικά καθεστώτα. Έχουμε την Περιφερειακή Συμφωνία ε, και όλα εκτός από τα όπλα για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες και το σύστημα γενικές, γενικευμένες προτιμήσεις συν για τις υπόλοιπες χώρες. Για το μέλλον των σχέσεων τονίζει τα εξή σημεία που θα περιληφθούν στην γνωμοδότηση. Πρώτον, στόχος μας πρέπει να έχουμε ένα αποτελεσματικό μετακοτονού πλαίσιο που να βασίζεται στο να αποδέχονται οι χώρες ε, της διατάξεις του και να είναι συμβατό με τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειάζεται επίσης ένα γενικό, μια συμφωνία γενικού πλαισίου που να στηρίξουν το δίκαιο εμπόριο και το βιώσιμο εμπόριο, ούτω ώστε να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και να μειωθεί η φτώχεια. Δεύτερον, όπως ξέρετε, η εταιρική σχέση Κοτονού είναι ένα πλαίσιο για να συζητηθούν τα εμπορικά θέματα με όλε τις 79 χώρε ΑΚΕ. Είναι σημαντικό να διατηρηθεί αυτό στην μελλοντική συμφωνία και να ενισχύσουμε την συνεργασία για εμπορικά και οικονομικά θέματα, για παράδειγμα για τις υπηρεσίες και η προσέγγιση μας να βασίζεται στην αξία που δημιουργείται, όπως προτείνεται στη στρατηγική εμπόριο για όλους, για να υπάρχει πιο υπεύθυνη εμπορική πολιτική. Επίσης, ε, ε, η περιφερειακή συνεργασία είναι πολύ σημαντική για το μέλλον των σχέσεων αυτών. Τρίτον, κατά τη γνώμη μου, η αναθεωρημένη συμφωνία πρέπει ε, να έχει αναθεωρημένους και βιώσιμους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι στόχοι για τα ουσιώδη στοιχεία πρέπει να παραμείνουν ούτως ώστε να συνεχίσουν να λειτουργούν οι συνθέσεις αυτές και μετά το 2020. Τέταρτον, επίσης τονίζω ότι πρέπει να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών. Αυτό είναι απαραίτητο για οποιαδήποτε συμφωνία. Και η παρακολούθηση της συνεργασίας είναι σημείο κλειδί, ιδιαίτερα όσον αφορά το εμπόριο και την ε, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Επιπλέον σημειώνω τη σημασία να συνεχιστεί αυτή η μεικτή ε, κοινοβουλευτική συνέλευση για να υπάρχει κοινοβουλευτική, κοινοβουλευτικός έλεγχος οποιασδήποτε συμφωνίας. Επίσης πρέπει να το συνδέσουμε όλο αυτό με τους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη της Αντίσα Μπέμπα και με τους στόχους για τη βοήθεια για την ανάπτυξη και για άλλη βοήθεια για τις χώρες αυτές για να αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και να αναπτύξουν τις περιφερειακές και παγκόσμιες αλυσίδες δημιουργίας αξίας. Ε, μας ευχαριστεί πάρα πολύ και προσβλέπει στη συνεργασία με τους κοιόδης για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο πρόεδρος Ντέιβιν. Και τώρα να δώσω το λόγο στους κοιόδης. Ο κύριος Ιένφελ πρώτα απ' όλα. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, από την πλευρά μου, το θέμα αυτό παρουσιάζει ορισμένες δυσχέρειες. Διότι αυτό που έχουμε πίσω μας είναι μια μακρά περίοδος ε, ευρείας συνεργασίας και στήριξης για τις χώρες ΑΚΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ευρεία συμμετοχή των κοινοτήτων. Έχουμε ακόμα μερικά χρόνια σε αυτό το πλαίσιο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να εργαστούμε για πώς θα συνεχιστεί με νέα μορφή αυτή η συμφωνία. Και νομίζω ότι τώρα είναι στιγμή να κάνουμε μια αξιολόγηση του πώς έχει λειτουργήσει. Η γνωμοδότηση αυτή Νομίζω ότι είναι πολύ αντικειμενική, ισορροπημένη, θίγει τα πιο σημαντικά θέματα όσον αφορά την εξολόγηση του παρελθόντος και του παρόντος. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πιο τολμηροί και να τονίσουμε τις ανάγκες μας για το μέλλον. Για την εφαρμογή της συμφωνίας με τις χώρες και τις λύσεις που πρέπει να εφαρμόσουμε για να... Ε, δεν μιλάω τώρα ειδικά για την ευρωμοδότηση, αλλά για τα αποτελέσματα της συμφωνίας μεταξύ των χρόνων και, και της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα. Εάν θα πρέπει οι χώρες αυτές να τις αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο. Είναι 80 χώρες από πολύ διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Πρέπει να συνεχίσουμε να τι αντιμετωπίζουμε ομοιόμορφα. Πιστεύω ότι για την περίοδο μετά το 2020 θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή μας την προσέγγιση. Και επίσης νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε ακριβώς την ε, αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, τι έχουμε επιτύχει μέχρι τώρα και δεν θα πρέπει, πιστεύω, να είμαστε επίοικείς με τους αυτούς μας. Οπότε, επειδή έχουμε ακόμη χρόνο, θα προτείνω ορισμένες ε, αλλαγές, θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες στην γνωμοδότηση, αλλά γενικά η γνωμοδότηση νομίζω ότι είναι καλή, αλλά νομίζω ότι χρειάζονται κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, κάποιες κρίσεις, κάποιες ε, συστάσεις που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ε, τα επόμενα χρόνια στη δουλειά μας. Τι συμφωνία θα επιδιώξουμε μετά το 2020. Αυτό είναι το θέμα. Ε, πρέπει να δούμε πιο συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε βοήθεια. Ίσως μάλιστα δεν θα πρέπει ούτε καν να χρησιμοποιούμε τον όρο βοήθεια. Πρέπει να μιλήσουμε για την συμμετοχή μας, την εμπλοκή μας στην κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη των χωρών αυτών. Ίσως έτσι θα πρέπει να το θέσουμε. Μέχρι τώρα θα έλεγα Συγγνώμη, ε, εννοώ ότι ε, η προσέγγιση που έχουμε έχει γίνει πλέον ε, πεπαλαιωμένη, αναχρονιστική. Εάν λοιπόν δεν τροποποιήσουμε τον τρόπο εμπλοκής μας, δεν θα ωφεληθούμε ούτε εκείνοι ούτε εμείς ούτε εμείς ως ε, πιθανοί επενδυτές στις ε, χώρες αυτές, διότι οι χώρες αυτές, όπως σας είπα, έχουν γίνει ήδη σημαντικοί μας εταίροι. Ε, τα, καθεστώτα, τα καθεστώτα τους είναι πιο φιλικά προς τις επιχειρήσεις και γίνονται σημαντικοί μας εταίροι και πολιτικοί και οικονομικοί. Πρέπει λοιπόν και αυτό να το λάβουμε υπόψη. Διότι θέλουμε φυσικά να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες και πρέπει να επιλέξουμε τα σωστά εργαλεία για να τις βοηθήσουμε. Ούτως ώστε να μην αισθανόμαστε απλώς ίσχυτη τη συνείδησή μα, αλλά να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα επιτόπου, θέσει εργασία, για παράδειγμα. Περισσότερη ευημερία, περισσότερη ανταγωνιστικότητα, τουλάχιστον σε περιφερειακές και υποπεριφερειακές αν όχι παγκόσμιες αγορές. Και τα μέσα που έχουμε αξιοποιήσει μέχρι τώρα, ναι, κοστίζουν πολλά, αλλά κατά τη γνώμη μου δεν είναι απόλυτα, απόλυτα αποτελεσματικά και πρέπει να το προσέξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η Έμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά που έχει ήδη γίνει πάνω σε αυτή τη γνωμοδότηση. Για μένα είναι πολύ σημαντικό το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ θα ε, βασιστεί στο εμπόριο και όχι στην ε, βοήθεια. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι χώρες θα έχουν πρόσβαση στο εμπόριο και ότι αυτό το εμπόριο θα τους δώσει την δυνατότητα ε, της, ε, να σταθούν στα πόδια τους και πιστεύω ότι το περιβάλλον ε, που έχει δημιουργηθεί στο Κοτονού δεν θα πρέπει να ολιστήσει προς ε, αναπτυξιακή βοήθεια, προς ε, συμπληρωματικές ενισχύσεις, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσει δυνατότητες διευκόλυνσης και ανάπτυξης του εμπορίου. Συμφωνώ στην, για την πλειοψηφία των σημείων της γνωμοδότησης. Θα ήθελα όμως να τονίσω το εξής, ότι ένα αποτελεσματικό πλαίσιο κοτονού θα πρέπει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το, τη διαφθορά και ε, μέσω της ε, διακυβέρνησης αλλά και ε, αυξάνοντας τη διαφάνεια. Πιστεύω ότι αυτό χρειάζεται έτσι ώστε να, δοθεί να αποκτήσει η εμπιστοσύνη η αγορά για να οδηγηθούμε στη διευκόλυνση του εμπορίου. Έπειτα, αμοιβαία απελευθέρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντική για να είναι αποτελεσματική, όμως πρέπει να συνοδεύεται με ανάπτυξη ικανοτήτων, με ανάπτυξη υποδομών και κυρίως με ε, ανάπτυξη δυνατοτήτων εξαγωγών. Γι' αυτό θεωρώ πως υπάρχει μία διαφορά μεταξύ μου και του εισηγητή για το νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα της βιώσιμης ανάπτυξης, για το κεφάλαιο αυτό. Δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες. Μου φαίνεται πολύ περίπλοκο αυτό που διαβάζω. Ίσως, βέβαια, γίνονται ήδη βήματα προς αυτό, αλλά θα μπορούσαμε ενδεχομένως να έχουμε ε, μια πιο απλή μορφή, έτσι ώστε να είναι και πιο ε, λειτουργική και να μπορέσουμε να αποκομίσουμε τα ωφέλη αυτής της συμφωνίας. Έχει γίνει ήδη πολλή δουλειά από τη Συμφωνία του Κοτονού και έπειτα και πιστεύω πως αυτή ε, η γνωμοδότηση μπορεί να βοηθήσει πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Χέλμουτ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και με τους συναδέλφους και με τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χαιρετίζω λοιπόν τις προσπάθειες του εισηγητή και θεωρώ το σχέδιο γνωμοδότησης μια πολύ καλή αφετηρία για να εξετάσουμε ε, από την προοπτική της Επιτροπής μας το μέλλον των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΚΕ. Και ερχόμενος από την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΠΟΕ, μπορώ να πω ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν, ε, συμμετέχουν και στον ΠΟΕ. Ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει εκεί. Βλέπουμε μία δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση των μελλοντικών συνθήκων. Από όλα τα 28 κράτη-μέλη, αλλά και από την πλευρά των χωρών ΑΚΕ. Η σκιώδη συγγήτρια, η κυρία Σάντσες, θα ήθελε να τονίσει ότι το ε, πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε είναι η Σύμβαση των ε, Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, διεθνείς συμβάσεις, το SDG και γενικότερα όλα αυτά θα πρέπει να συνεισφέρουν σε ένα πλαίσιο που θα ευνοεί την ανάπτυξη της δημοκρατίας αλλά και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και εμείς από την QNGL θέλουμε να τονιστεί ότι πρέπει να, να δοθεί έμφαση σε συγκεκριμένα σημεία για το μέλλον, δηλαδή ότι η διαδικασία του κοτονού θα έπρεπε, θα πρέπει μάλλον να δώσει ένα ισορροπημένο ε, πλαίσιο όπου οι εταίροι θα συζητούν για θέματα δίκαιου εμπορίου επίσης ώρες και αυτές οι σχέσεις θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι έχουν και ε, προβλήματα εκτός από πλεονεκτήματα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να συνδέσουμε και ε, το εμπόριο με αυτά τα προβλήματα και πώς αυτά θα ξεπεραστούν. Επίσης, να τονίσουμε την επιθυμία μας για νομικά δεσμευτικά μέσα, για ε, την ανάληψη ευθυνών από τον ιδιωτικό τομέα και, από τη, και για την καταπολέμηση της ε, διεθνούς ατιμορρησίας. Είναι, νομίζω, μία οριζόντια υποχρέωση για να, δούμε δηλαδή το, τις διασυνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στο εμπόριο με αυτές τις χώρες και σε μας. Είναι εξάλλου θέμα αμοιβαίου σεβασμού. Αυτό υπάρχει και ε, στον στόχο αριθμό 15 για το καθήκον των χωρών να ε, ασκούν. Είναι λοιπόν ο αναπτυξιακός στόχος 15, ο οποίος αναφέρει αυτήν την υποχρέωση βιωσιμότητα του χρέους, θέματα συνεργασίας ε, τα οποία θα καταπολεμήσουν τις παράνομες ροές κεφαλαίου. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω ότι στη Γενέβη συζητήθηκε και κάτι άλλο σημαντικό. Πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειες καταπολέμησης της διαφθοράς. Αυτό αναφέρθηκε από πολλούς συμμετέχοντες. Και αναφέρθηκαν επίσης ε, τα θέματα της ε, δημογραφικής αλλαγής σε πολλές περιοχές. Έχουμε όλοι κοινέ αξίες και κοινού στόχους, γι' αυτό λοιπόν η ομάδα μας θα υποβάλει τις σχετικές τροπολογίες και ελπίζουμε σε μια επικοδομητική συνεργασία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρούας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ να πω κάποια πράγματα. Βέβαια, τα περισσότερα έχουν ήδη υποθεί, αλλά δράτω με τις ευκαιρίες να τονίσω τη σημασία της εταιρικής σχέσης και της εργασίας που έχει κάνει ο εισηγητής. Διότι νομίζω ότι είναι πολύ ισορροπημένη. Έχω κάποιες τροπολογίες να καταθέσω, οι οποίες όμως δεν αντιβαίνουν στις προθέσεις της έκθεσης. Όπως είπα, είναι ιδιαίτερα ισορροπημένοι, αλλά είναι κάποια στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Καταρχάς, οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Να τονίσω ότι όχι μόνο ε, υπάρχουν νέες προκλήσεις που αναδύονται, και αυτό πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση, αλλά ναι. υπάρχει και το κομμάτι της πάταξης της φτώχειας. Πρέπει να μπορέσουμε να μιλήσουμε πλέον για την πλήρη πάταξη της φτώχειας, ε, γιατί στην έκθεση λέει απλώς για τη μείωση της ε, φτώχειας. Επίσης, η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Έχουμε μιλήσει για την ευθύνη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και οι εταιρείε πρέπει να αναφερθούν, θεωρώ. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Όταν μιλάμε για αξίες, πρέπει να αναφέρουμε την βιώσιμη ανάπτυξη. Αναφέραμε την ανάπτυξη, αλλά όχι τη βιώσιμη ανάπτυξη στην έκθεση και θα προτείνω μία τροπολογία σε αυτό το πνεύμα. η δουλειά του Πέτρο Σίλβα Περέιρα είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά στη μεικτή κοινοβουλευτική ε, συνέλευση και την προηγούμενη συζήτηση που έχει γίνει για αυτό το θέμα. Αδειμονούμε για αυτή την εταιρική σχέση, όμως είναι πολύ σημαντικό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ταυτόχρονα να σκεφτεί όλα αυτά τα ζητήματα. Η μεικτή κοινοβουλευτική συνέλευση είναι ένα σώμα μεγάλη σημασία ε, έχει μεγάλη, ένα σημαντικό ρόλο να παίξει στις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είναι λοιπόν μια εκθέση πολύ σημαντική και μαζί με τις ε, τροπολογίες που θα καταθέσω θα είναι πολύ ε, πιο σημαντική νομίζω. Ευχαριστώ. Και Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, ε, έχουμε εδώ δύο εκπροσώπους της Επιτροπής, δύο εκπροσώπους από δύο διαφορετικές γενικές διευθύνσεις. Θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις τους. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Δεν χρειάζεται να πω ότι οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών ΑΚΕ είναι παλιές. Η Συμφωνία Κοτονού ήταν μοναδική λόγω του δεσμευτικού νομικά χαρακτήρα της, του περιεχομένου της, των παραγόντων που ε, παίζουν ρόλο σε αυτή. Έχουμε κάνει μεγάλη δουλειά σχετικά με τα προηγούμενα και την τρέχουσα συμφωνία που θα καταλήξει τον Ιούλιο. Νομίζω επίσης ότι ε, με αυτά που κάνουμε θα μπορέσουμε να πατάξουμε τη φτώχεια, να φέρουμε ε, ειρήνη και ασφάλεια, αλλά πάντοτε υπάρχει περιθώριο για βελτιώσεις. Τώρα, για τη μελλοντική σχέση, πώς πρέπει να αναπτυχθεί. Πρέπει να βασίζεται στα κοινά συμφέροντα φυσικά, ξεκινώντας με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κοινό έδαφος. Ε, αυτό, βέβαια, πάει πέρα από την ανάπτυξη και στο Συμφωνία Κοτονού υπήρχε αυτό το κομμάτι, διότι μιλάμε για ίσους εταίρους. Υπάρχουν ζητήματα που είναι παγκόσμια εμβέλειας, πολιτικά, ασφάλεια των επιχειρήσεων, εμπόριο, μετανάστευση. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ κέρια. Πρέπει να μπουν στο πλαίσιο το καινούριο, διότι δεν είναι τα πλάγματα τα ίδια ε, όπως ήταν το 2000. Υπάρχουν πολλές αλλαγές. Επίσης έχουμε την Ατζέντα 2030 και τους στόχους δημο... βιώσιμης ανάπτυξης. Πρέπει και αυτά να μπουν στο παιχνίδι. Ε, υπάρχει μια ατζέντα για τους στόχους αυτούς και θα προσαρμοστεί και η Ευρωπαϊκή Συνένωση για την Ανάπτυξη, Συνένεση για την Ανάπτυξη σε σχέση με αυτό το θέμα. Αφού αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα το κάνουμε. Η επικουρικότητα και η συμπληρωματικότητα είναι πολύ σημαντικές αρχές. Σε, ε, ε, έχουμε το εθνικό, το περιφερειακό, υποπεριφερειακό ε, επίπεδο. πρέπει να δούμε πώς ε, θα προχωρήσουμε, ποιο επίπεδο θα ακολουθήσουμε. Ίσως το εθνικό επίπεδο να παραμένει το πιο αποδοτικό. Έχουμε δει τα εργαλεία, μαθαίνουμε από τα μαθήματα που έχουμε ήδη λάβει βάσει της εμπειρίας μας και θα δούμε και ποιοι θα είναι οι συμμετέχοντες σε αυτή την εταιρική σχέση, ποιοι παράγοντες θα εμπλακούν η κοινωνία φυσικά και ο ιδιωτικός τομέας. Θα αποτελέσουν αυτά λοιπόν τα δομικά στοιχεία για την πρόταση που θα κατατεθεί προ τα τέλη του έτου. Ευχαριστώ. Και ο συνάδελφο, σα παρακαλώ. Ή συνάδελφο. Καλησπέρα σα. Θα είμαι σύντομη. Θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με τα EPA τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης δηλαδή. Είναι ζωτικό λοιπόν να μείνουν οι θεμελιώδεις ρήτρε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό θέλουμε οπωσδήποτε να επιτύχουμε σε αυτές τις συμφωνίες. Αυτό είναι το ένα. Για κάτι άλλο στην γνωμοδότηση είναι η συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. Σήμερα το πρωί συζητήσατε μια συγκεκριμένη τέτοια σχέση και ξέρετε ότι είναι βασικό στοιχείο οποιασδήποτε τέτοια συμφωνία. Ακόμη λοιπόν και μετά την λήξη της συμφωνίας Κοτονού θα εξακολουθούμε να το έχουμε στο κέντρο της προσοχής μας. Ευχαριστώ πολύ. David, θέλεις να προσθέσεις τίποτα? Ναι, να τονίσω ότι η γνώμη του Πέντρο ε, δεν θα πρέπει να ε, συγχαίεται με την έκθεση. Η γνωμοδότηση αφορά μόνο την πλευρά του εμπορίου. Και ο συντάκτης της ασχολείται μόνο με τα εμπορικά θέματα. Για τη βοήθεια, για παράδειγμα, δεν έκανε ευρύτερα σχόλια, αλλά ζήτησε να ενισχυθεί η βοήθεια για το εμπόριο που νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να το ζητήσει η Επιτροπή μα και είναι και σωστή στρατηγική, ούτω ώστε οι χώρες της ΑΚΕ να μπορέσουν να ενταχθούν στο παγκόσμιο σύστημα εμπορικών συναλλαγών. Επίσης, τονίζει ιδιαίτερα κάτι που μας ενδιαφέρει, ότι θα πρέπει να τις ε, αντιμετωπίσουμε ενιαία Ορισμένοι λένε ότι θα έπρεπε να χωρίσουμε τις χώρες ΑΚΕ σε τρία τμήματα, αλλά εκείνο θεωρεί ότι πρέπει να είναι μια ενιαία εταιρική σχέση. Και παραλαμβάνω αυτό που είπα στην αρχή, υπάρχουν τρεις πυλώνες στη σχέση μας. Το εμπόριο είναι ένας πυλώνας. Ό,τι και αν γίνει στην αξιολόγηση, το εμπόριο πρέπει να παραμείνει πυλώνας. Και ίσως θα έπρεπε να γίνει ο πυλώνας της σχέσης μας με τις χώρες ΑΚΕ. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης θα γίνει 13-14 Ιουλίου με βάση το πρόγραμμα προθεσμία για τροπολογίες 21 Ιουνίου 18 6 ώρα το απόγευμα και θα εξετάσουμε τις τροπολογίες την 31 Ιουνίου λέει ο Πρόεδρος στη συνεδρία της Επιτροπής μας Εδώ λέει 31, αλλά δεν μπορεί να είναι 31, είναι 30. 30 Ιουνίου. Αγαπητοί συνάδελφοι. Υπάρχει μια εξαιρετική κατάσταση. Τελειώσαμε νωρίτερα από ό,τι είχαμε προγραμματίσει. Εντελώς ασυνήθιστο. Η ακρόασή μας αρχίζει στις 4.30. Ε, Έχουμε λοιπόν μια διακοπή 14 λεπτών. Και θα αρχίσουμε αρχηγός, ακριβώς 4 και 30. Παρακαλώ μόνο καφέ, μόνο καφέ και μετά να ξανάρθετε.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 So, ladies and gentlemen, please take your seats. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Mr. Leeds. So, ladies and gentlemen, dear... Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω σε αυτή τη δημόσια ακρόαση που διοργάνωσε η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Σήμερα εστιάζουμε στην Ευρωπαϊκή Εμπορική Πολιτική στα πλαίσια της ε, Διεθνούς Αλυσίδας Αξιών. Μένοντας πιστή στην αρχή της βιωσιμότητας και πώς μπορούμε να εντάξουμε τη βιωσιμότητα στην παγκόσμια Αλυσίδα αξιών. Για μένα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι το εμπόριο έχει αλλάξει τα τελευταία 20 χρόνια. Και μάλιστα ε, νομίζω πως έχει αλλάξει τόσο ώστε να μην μπορεί να παρακολουθήσει ούτε ο Ντέιβιντ Ρικάρντο τις εξελίξεις. πλέον δεν ανταλλάσσουμε και δεν εμπορευόμαστε προϊόντα, αλλά και διάφορα διάμεσα στάδια. Υπάρχει δηλαδή μία λυσίδα αξιών που φτάνει στο 75% της, ε, του παγκόσμιου εμπορίου. Η εμπορική πολιτική, για να εκτιμηθεί σωστά, είναι πολύ σημαντικό είτε να υπάρχουν εμπορικές συμφωνίες, είτε να κοιτάξουμε μεγαλύτερη προσοχή την παγκόσμια λυσίδα αξιών. Σήμερα το βράδυ θα γίνει τριμερής διάλογος με το Συμβούλιο για την Ομοθεσία σχετικά με τα ορυκτά από εμπόλεμες ζώνες. Είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην παγκόσμια λυσίδα αξιών, αρχίζοντας από το πιο απλό και φτάνοντας μέχρι, μέχρι ένα smartphone το οποίο είναι και ένα πολύ καλό παράδειγμα της παγκόσμιας αλυσίδας αξιών. Ένα τέτοιο κινητό τηλέφωνο περιέχει διάφορα πλαστικά, διάφορα μέταλλα, τα οποία διανύουν τεράστιες αποστάσεις. Μέχρι 32.000 χιλιόμετρα έχουν διανύσει όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για να φτιαχτεί ένα τέτοιο τηλέφωνο. Και διασχίζουν περίπου 100 σύνορα μέχρι να φτάσουν στην διαδικασία κατασκευής. Αυτό δηλαδή είναι ε, ένα δείγμα του πόσο σημαντική είναι η αλυσίδα αξιών. Μας ζητείτε λογοδοσία και από τις επιχειρήσεις και από τους νομοθέτες σε αυτήν την παγκόσμια αλυσίδα αξιών. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που σήμερα μπορούμε να το συζητήσουμε με εμπειρογνώμονες και με συναδέλφους από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Δύο αλυσίδες αξιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Ο τομέας της ένδυσης Η τραγωδία του Ουράνα Πλάζα έχει τώρα τρία χρόνια που έχει συμβεί και δεν είμαι πεπισμένος ότι έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε να υπάρχει εγγύηση ότι η αλυσίδα εφοδιασμού θα είναι δίκαιοι στον τομέα της ένδυσης. Νομίζω πως η Επιτροπή Ανάπτυξης και όλας έχει μια ενδιάμεση έκθεση την οποία θα στηρίξουμε και εμείς. Από την άλλη, πολύ σημαντικός τομέας είναι ο τομέας των τροφίμων και της γεωργίας. Και εδώ Πρέπει να συζητηθεί το θέμα της βιωσιμότητας στην παγκόσμια λυσίδα αξιών, ιδιαίτερα για το εργατικό δυναμικό. Είναι λοιπόν σημαντικά ζητήματα αυτά. Και στη σύνοδο των ε, G7 συζητήθηκε το θέμα της διαφάνειας στην παγκόσμια λυσίδα αξιών. Πιστεύω πως ε, δεν συζητήθηκε παρκώς και θα έπρεπε να εμβαθύνουμε ίσως. Αυτό θα συζητήσουμε και σήμερα. Εάν δηλαδή οι κανόνες του εμπορίου και οι εμπορικές πρακτικές θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα και το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι θα χαρακτηρίζονται από βιωσιμότητα. Έχουμε μαζί μας δύο διακεκριμένους εμπειρογνώμονες. Ο πρώτος ομιλητής από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Σάντρα Γκαλίνα. Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εμπειρογνώμων λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σας δίνω αμέσως το λόγο για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Με χαρά μου βρίσκομαι σήμερα εδώ. Θα ήθελα να πω κατευθείαν στο ζητούμενο. Οι παγκόσμιε αλυσίδε αξία δεν θα πρέπει να γίνουν ένα μέσο για να γίνουν πιο αδιαφανεί, ε, για να μην γνωρίζουμε πώ ακριβώ παράγονται τα αγαθά. Υπάρχουν πολλέ πτυχέ αυτό και που αφορούν όλους, όχι μόνο τους μεγάλους παραγωγούς, μεγάλες αλυσίδε, αλλά και τους μικρούς παραγωγούς. Θα έπρεπε ίσω να γνωρίζουμε ότι η διαφάνεια που απαιτούν οι καταναλωτές δεν είναι ε, κάτι ασήμαντο, δεν είναι ένα ακόμα κομμάτι της εταιρική ευθύ, κοινωνικής Όχι. Αφορά όλους. Καταρχάς, να σα πω ότι είναι πολύπλοκο το ζήτημα και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντε που συνεισφέρουν. Για να καταλάβουμε τις διαστάσεις θα σας πω το εξής. Υπάρχει εξωτερική διάσταση και ως ε, εκπρόσωπος της ε, ΓΔ Εμπορίου Είμαι μέρος αυτής. Εκπροσωπώ λοιπόν την εξωτερική διάσταση, αλλά και έχω σε ένα συνάδελφο δίπλα από τη ΓΔ η οποία Γενική Διεύθυνση έχει πολιτικές που ε, αφορούν τις υπεύθυνε εμπορικές πρακτικές. Πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη εσωτερική εγχώρια διάσταση, η οποία είναι αρμοδιότητα της ε, γαμα-δέλτα-γκρόου. Grow. Πολλές φορές υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνο γιατί και ποιος κάνει τι. Πολλοί δεν ξέρουν. Και το λέω αυτό διότι υπάρχουν ολόκληροι τομείς πολιτικής που ε, επηρεάζονται και πολλές φορές λείπουν ολόκληρα κομμάτια πολιτικής ε, τα οποία αφορούν εξωτερική πολιτική, την εξωτερική διάσταση, η οποία επίσης παίζει ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ το θέμα και η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, την οποία προσπαθώ να εκπροσωπήσω, έχει ορισμένα ε, μέσα στην εργαλειοθήκη της και τώρα θα σταθώ και στο θέμα του Μπαγκλαντές που ανέφερε και ο Πρόεδρος, γιατί νομίζω πως έχουμε πολλά σημαντικά να πούμε. Όπως είπα, είναι πολύπλοκο το σύστημα. Εμείς ως ε, ΓΑΜΑ Εμπορίου προσπαθούμε να ε, δραστηριοποιούμαστε όχι μόνο σε πολυμερές πλαίσια, αλλά και σε μονομερές. Έχουμε το GSP ε, Plus, ο συνάδελφος ο Νίκος είναι δίπλα μου υπεύθυνο γι' αυτό. Υπάρχει ε, η πολιτική για τις υπεύθυνε ε, επιχειρηματικές πρακτικές, οι οποίες αφορούν βασικά εργασιακά πρότυπα. Αυτή λοιπόν είναι η μονομερής διάσταση, διεμερής τώρα διάσταση. Υπάρχουν, όπως λέμε, κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, σχετικές διατάξεις. Σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν, όμως είναι η αφετηρία μιας δράσης. Επίσης, η δραστηριοποίηση σε πολυμερές πλαίσιο. Εδώ πρέπει να βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε την παρουσία μας διότι θεωρώ πως ε, η Ευρώπη μόνη της δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την διαδικασία. Πρέπει να κατευθυνθούμε περισσότερο στους ε, διεθνείς οργανισμούς, να στρέψουμε το βλέμμα εκεί και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Νομίζω πως υπάρχει και ένας ομιλητής ε, στο πάνελ από τον ΩΣΑ και νομίζω πως θα σας αναφέρει όλες τις πρωτοβουλίες τις οποίες στηρίζει και χωρική Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τομέα της ένδυσης και της υπόδησης, Έτσι ώστε να αποφεύγεται το κοινωνικό ντάμπινγκ. Και πρόσφατα στο Σιάτλ απέρριψαν και ήταν κάθετα κατά των δικών μας προτάσεων. Τώρα, μπορώ να πω ότι εμείς προσπαθούμε να καινοτομήσουμε. Έχουμε αυτά τα ορυκτά από εμπόλεμες περιοχές, όπως είπατε. Υπάρχει ο υποχρεωτικός ή ο προαιρετικός χαρακτήρας, όμως σε κάθε περίπτωση και στις δύο μάλλον περιπτώσεις πρέπει να γίνονται σεβαστά αυτά τα πρότυπα. Ε, υπάρχει το σύμφωνο του Μπαγκλαντές. Ίσως έχετε διαβάσει τα πρόσφατα σχετικά έγγραφα. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή ως Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούμε να δώσουμε ε, έμφαση και να στρέψουμε την προσοχή στην ασφάλεια στον χώρο εργασίας. Ε, χρειάζεται όμως να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες. Αρχίσαμε δηλαδή ε, τη συζήτηση με την κυβέρνηση του Μπαγκλαντές, τώρα χρειάζεται όμως να εμβαθύνουμε. Να εμβαθύνουμε σε κάτι το οποίο δεν παραμελήσαμε, αλλά προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε με λεπτότητα, ακριβώς γιατί είναι ευαίσθητο ζήτημα. Τι κάνουμε τώρα, προσαρμόζουμε την προσέγγιση σε αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Δηλαδή, ε, οι συνταγές ε, του πώς γίνεται ε, δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολεί εσάς. Εσείς είστε η πολιτική εγκέφαλοι πίσω από αυτό. Έχετε άλλες αρμοδιότητες και δυνατότητες. Στι ε, Παγκόσμιες ημέρε ο Επίτροπος το ανέφερε και ότι εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να βοηθήσουμε, να ενισχύσουμε αυτήν την άποψη του εμπορίου, διότι πολλά προϊόντα έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, PPM στα λέμε αυτά, στον ε, Τώρα, χρειάζεται να χτίσουμε εμπιστοσύνη. Πολλές φορές χρειάζεται πολιτική παρέμβαση γι' αυτό. Δεν επαρκούν οι τεχνοκράτες όπως εγώ. Δεν μπορούμε να πείσουμε κυβερνήσεις. Ο ιδιωτικός τομέας πρώτα-πρώτα πρέπει να διαπιστώσει ότι υπάρχει μία αγορά και χρειάζεται η αγορά αυτή να έχει από πίσω της μία κυβέρνηση που να τη στηρίζει. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το κάνει αυτό από μόνη της. Όχι. Χρειάζεται η πολιτική πίεση όπως και σε άλλες περιπτώσεις, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, που πιέζουν για να αλλάξουν καταστάσεις. Χρειάζεται επίσης χρόνος για να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Ενδεχομένως είδατε τα αποτελέσματα του συνεδρίου της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας. Προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε ένα, ένα δρόμο και να πω εδώ ότι αυτή τη στιγμή 9 εκατομμύρια έχουν ε, ανατεθεί στη δημιουργία ευαισθητοποίησης για υπεύθυνες εμπορικές πρακτικές στην Ασία. Και θα Σα αναφέρω ακριβώς τι κάνουμε, γιατί θεωρώ πως είναι σημαντική πρωτοβουλία. Συνοψίζοντα λοιπόν, ε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη, να δημιουργήσουμε αμοιβαιότητα. Δεν πρέπει μόνο εμεί να κάνουμε προτάσεις, πρέπει και οι άλλοι να τις δέχονται. Προσπαθούμε να κάνουμε μια διαλογή για να δούμε τις πιο σημαντικέ ε, δράσει μονομερείς και διμερείς προσεγγίσεις λειτουργούν καλύτερα από τις πολυμερείς και έπειτα κοιτάζουμε πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις ιδέες μας για ε, την ε, ευθύνη και για την υπευθυνότητα. Και τέλος, ε, ο ρόλος της δράσης είναι σε εσά τα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω τώρα την Προεδρία στον ε, συνάδελφό μου, τον κύριο Κούλογλου. Αντιπρόεδρο, ζητώ συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος, ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης, που θα είναι και ο συμπρόεδρος στο πρώτο πάνελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι, δικές, οι επιτροπές μας είχαν πρόσφατα μια κοινή συζήτηση για μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καιρό περιμέναμε για την διαχείριση της αλυσίδας αφοδιασμού του τομέα των ενδυμάτων, της ένδυσης. Με πολύ χαρά σήμερα θα συνεχίσω την συζήτηση για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Δεν ξέρω πόσοι από εμά ακόμα θυμόμαστε πόσοι πέθαναν το ατύχημα του Ράνα Πλάζα. Θυμάται κανείς πόσοι. Εκτός μικροφώνου, ακριβώς 1138 πέθαναν. Όμως δεν θυμάται πολλοί ε, κόσμος αυτή την τεράστια τραγωδία. Τρία χρόνια μετά η Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ προχωρά με μία προσέγγιση που εμπλέκει όλους τους ενδιαφερόμενους για να μπορέσει να προωθήσει μια πιο υπεύθυνη στάση στον τομέα της ένδυσης, να προωθήσει τα ανθρώπινα ε, εργασιακά δικαιώματα και κάθε είδους ε, τέτοιο δικαίωμα σε αυτές τις χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί προορισμό για αυτές ε, τις ε, βιομηχανίες και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν πολιτικές και δράσεις επιγόντως σε αυτούς τους τομείς. Όπως αναγνωρίζει το Συμβούλιο στα πρόσφατα συμπεράσματά του του Μαΐου 2016 για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπεύθυνε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας και αναφέρω τα λόγια τους. Ε, αυτό το θέμα έχει πολύ μεγάλη σημασία ε, μέσα στα πλαίσια ε, των τρέχοντων τρέχουσων εξελίσεων καθώς οι χώρες οι αναπτυσσόμενες συνεχώς αλλάζουν ε, και απαιτείται μεγαλύτερη προώθηση της ανάπτυξης για τις πιο ευαίσθητες χώρες. Οι παγκόσμιες αλυσίδες αξίας λοιπόν μπαίνουν στο προσκήνιο, διότι υπάρχουν είναι σκάνδαλο πόσο τραγικές είναι οι συνθήκες εργασίας, ε, όπως ήταν ε, οι συνθήκες στο Ράνα όπου κατέρευσε το εργοστάσιο. Έχουμε συνεχώς προβλήματα διαρθρωτικού επίπεδου στην βιομηχανία. Δεν υπάρχει ε, ένας ε, μισθός ε, που να μπορεί κανείς να επιβιώσει, εργασία διαπόστασης. Υπάρχουν τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπάρχει περιβαλλοντική ρήπανση και διάφορα τέτοια προβλήματα στις χώρες με τα χαμηλότερα ημερομίσθια. Οι περισσότερες εισαγωγές ε, ενδυμάτων γίνονται από την Ασία. Συνήθως είναι οι γυναίκες που εργάζονται στον τομέα αυτό. Στον Μπαγκλοντές μια γυναίκα μπορεί να βγάζει 60 ευρώ το μήνα. Τόσο λίγο. Δεν μπορεί να ζήσει κανείς με αυτά τα χρήματα. Σε χώρες γειτονικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, έχουμε παιδιά που δουλεύουν. Πολλοί κακές συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς, αυτά είναι κοινό, φαινόμενο. Και τώρα έχουμε και τους πρόσφυγες που προστίθενται σε αυτό. Ε, έτσι λοιπόν δεν υπάρχει συμμόρφωση ούτε ηθική, ούτε νομική. Ακόμα και μετά από αυτές τις καταστροφές και την κριτική που δέχτηκαν οι χώρες αυτές σε δημόσιο επίπεδο. Η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να βοηθήσει στο να ενισχύσουμε την υπεύθυνη στάση των επιχειρήσεων στον τομέα των, ε, της ένδυσης. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε κοινέ πρωτοβουλίες, ε, να βρούμε τις συνέργειες και φυσικά να μην εξαιρέσουμε τα νομοθετικά μέτρα. Εδώ πρέπει να κάνουμε και έναν παραλληλισμό με την ευρωπαϊκή ε, δράση για τη βελτίωση των ε, πρακτικών, επιχειρηματικών πρακτικών και την αύξηση της λογοδοσίας ε, στον τομέα της εξόριξης και των μεταλλίων, για παράδειγμα. Αυτές οι βιομηχανίες μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και, είμαστε και έχουμε μεγάλη ευθύνη. Όχι μόνο ως προς τους εργαζόμενους, στις χώρες αυτές με τις οποίες εμπορευόμαστε, αλλά και απέναντι στους καταναλωτές στις χώρες μας. Προσκαλώ λοιπόν ε, τους ομιλητές, ξεκινώντας με τον ε, Σέρι Στέφενσον, που είναι βασικός συνεργάτης του Διεθνούς Κέντρου για, την, ε, για το και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, να μας μιλήσει για το θέμα. Ή κυρία Στέφενσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ε, πρόσκληση να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Θα κάνω μια γενικότερη επισκόπηση ε, σχετικά με το θέμα της διακυβέρνησης και των παγκοσμίων ε, αλυσίδων αξίας και τι σημαίνει αυτό για το σύστημα. Σήμερα είμαστε σε μια οικονομία στην οποία οι επενδύσεις ηγούνται έχουμε ότι τα τρία τέταρτα των υπηρεσιών ε, είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε λοιπόν ε, επιχειρήσεις που δρούν σε αυτό το πεδίο. Οι περισσότερες ε, κυβερνήσεις θέλουν οι εταιρείες τους να έχουν αυτές τις δομές παγκόσμια αλυσίδα αξία, γιατί έτσι θα έχουν και μεγαλύτερη και δυναμική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, έχει γίνει μια έρευνα που δείχνει ότι οι εταιρείε, οι χώρες αυτές που ενσωμάτωσαν αυτές τις δομές ε, μπόρεσαν να αναπτύξουν την οικονομία τους 2% πιο γρήγορα την περασμένη δεκαετία από τις υπόλοιπε. Δυστυχώ, οι αναπτυσσόμενε χώρες στην παγκόσμια οικονομία δεν είναι κοντά στα κέντρα αυτών των ε, δραστηριοτήτων ε, που βρίσκονται σε 40 με 50 χώρες στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Ανατολική Ασία. Ε, έχουμε λοιπόν διαφορετικούς ε, παράγοντες. Οι αλυσίδες αξίας οργανώνουν την παραγωγή χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα σύνορα. Θα πρέπει κανείς λοιπόν να λάβει μέρος σε αυτές τις αλυσίδες για να μπορεί να προωθήσει τις δεξιότητες και το εμπόριο στη χώρα τους. Οι αλυσίδε αξίας είναι ένας νέος τρόπος ε, ε, διεξαγωγής του παγκοσμίου εμπορίου. Ε, έχουμε κανόνες και κανονιστικά πλαίσια. Αυτό σημαίνει ότι η διακυβέρνηση αυτών των αλυσίδων λαμβάνει υπόψη διαφορετική οπτική γωνία. Ποιο λοιπόν διακυβερνά αυτέ τι αλυσίδε εξαρτάται από το ποιο απαντά στην ερώτηση. Διότι μπορούμε να έχουμε τρεις, τρία επίπεδα τις εταιρείε, τις χώρες και το Διεθνές Σύστημα Εμπορίου. Ας εξετάσουμε το καθένα χωριστά. Σε επίπεδο εταιριών, η διαχείριση εκεί είναι ξεκάθαρη. Έχει να κάνει με το πώς οργανώνονται οι δραστηριότητες στο όλο δίκτυο των επιχειρήσεων. Ενισχύονται οι παράμετροι με τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο. Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο, λοιπόν, κυρίως οι πολυεθνικές είναι αυτές που διακυβερνούν ε, τις επενδύσεις, το outsourcing και όλες αυτές τις δραστηριότητες ε, της αλυσίδας. Ε, ε, αυτές είναι τα κίνητρα. Αυτοί που συμμετέχουν στις αλυσίδες θέλουν να ενισχύσουν το κέρδος τους σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Και πώς τοποθετούν τον εαυτό τους σε μια τέτοια αλυσίδα. Αυτό πάλι εξαρτάται από το ποιος θέτει το ερώτημα. Έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν τις επιλογές μέσω της εφαρμογής συμβάσεων στις διάφορες χώρες. Έτσι λοιπόν ε, πολλές φορές γίνονται κάποια παζάρια μεταξύ των κρατών και των τοπικών επιχειρήσεων. Ο στόχος των επιχειρήσεων λοιπόν ε, είναι να δημιουργηθεί όσο πιο αποτελεσματική παραγωγή. Το βασικό ερώτημα σε αυτό το επίπεδο είναι πώς όμως μοιράζονται τα ωφέλη μεταξύ των μεγάλων εταιριών και των μικρομεσαίων ε, συμμετεχόντων στο δίκτυο αυτής της αλυσίδας. Στο επίπεδο τώρα του κράτους έθνους, η κάθε κυρίαρχη κυβέρνηση θέλει να διακυβερνήσει αυτή την αλυσίδα. Είναι μια πρόκληση για να δημιουργήσει μια σειρά πολιτικών που θα τις επιτρέψουν να λάβει μέρος σε αυτές τις διαδικασίες. Η διαχείριση σε αυτό το επίπεδο βασίζεται ε, στην ε, ε, πρόθεση των χωρών να έχουν μια καλή ευνοϊκή θέση στην παγκόσμια αγορά. Είναι δραστηριότητες που θα ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την τεχνολογία, τις δεξιότητες και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολλοί αναλυτές έχουν πει ότι η ατζέντα κυρίως πρέπει να είναι κρατική, τοπική για να μπορεί μια χώρα επιτυχημένα να συμμετέχει σε τέτοιες αλυσίδε αξίας θα πρέπει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις. Υπάρχουν πολλοί τομείς ε, που άπτονται αυτού του θέματος. Ε, μια φιλελεύθερη πολιτική είναι σημαντικό κομμάτι. Οι ανοιχτές αγορές ε, δεν μπορούν όμως να είναι αποτελεσματικές χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό που θα δώσει τη δική του, ε, θα βάλει το δικό του λιθαράκι. Είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις πολιτικές να δίνονται ανταγωνιστικές, μια πιο ανταγωνιστική διάσταση, να είναι η κυβερνητική τα θεσμικά όργανα στις κυβερνήσεις ε, μη διεφθαρμένα και να υπάρχει μια καλή υποδομή που θα συνδέει τις χώρες με τον υπόλοιπο κόσμο, να είναι καλή διαχείριση των ε, τελωνίων και των συνόρων και φυσικά να, οι τοπικοί κανονισμοί να μην ε, έχουν διακρίσεις. Στο διεθνές τώρα σύστημα εμπορίου δεν έχουμε διερευνήσει πολύ τα πράγματα. Δεν έχει σημασία το μεμονωμένο επίπεδο. Έχουμε ένα ευρύτερο επίπεδο που έχει να κάνει με διάφορους ε, ε, εταίρους στο, στην εμπορική αλυσίδα. Ε, υπάρχει βέβαια εδώ ένα κενό διακυβέρνησης που έχει αφήσει ο ΠΟΕ λόγω της μεγάλης τεμονής στην ατζέντα του κυγύρου της Ντόχα. Και έτσι δεν υπάρχει συντονισμός. Έχουμε κάποιες ε, τοπικές συμφωνίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει μια πειθαρχία για τα μέλη της. Έχουμε βέβαια κάποιες άλλες ε, διαπραγματεύσεις σε ευρύτερο επίπεδο όπως το TTIP, το RCEP και το TPP ε, που θα επηρεάσουν σε συστημικό επίπεδο τις αλυσίδες. Ξέρουμε ότι αυτό το κενό έχει δημιουργηθεί γιατί οι κανόνες του ΠΟΕ είναι παροχημένοι. Πριν από 20 χρόνια ήταν ότι ήταν μια αναδυόμενη τεχνολογία μόλις είχε εμφανιστεί ο παγκόσμιος ε, ιστός. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει κάλυψη, δεν υπάρχουν οι βασικοί τομείς στον ΠΟΕ, υπάρχει ένα κενό ε, δεν υπάρχουν κανόνες ας πούμε για τις επενδύσεις, τον ανταγωνισμό, το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό εμπόριο και στο ΠΟΕ δεν υπάρχει ένα φόρουμ που θα επιτρέπει στα μέλη του να συζητούν όλα τα θέματα έτσι ώστε οι εταιρείες να μπορούν να εμπλέκονται σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και να συζητούν για αυτά. Να καταλήξω λοιπόν, επειδή η διαχείριση των ε, αλυσίδων αξίας ε, είναι ένα θέμα που μπορεί να δει κανείς από διάφορες οπτικές γωνίες, ε, πρέπει όλοι να συμμετέχουν στο διάλογο. Οι εταιρείες, τα κράτη, τα κράτη μπορεί ε, να έχουν αντικρώμενα συμφέροντα ε, με τους υπόλοιπους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Έτσι λοιπόν, αν ο ΠΟΕ δεν αναλάβει δράση με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, αν θα έχουμε όλο και περισσότερες περιφερειακές συμφωνίες που θα καλύπτουν το κενό αυτής της διακυβέρνησης και θα παραμένουμε με την ίδια κατάσταση. Ευχαριστώ. So we got... Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε λοιπόν το συνολικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ένα σημαντικός κλάδος. Οι επιχειρήσεις. Έχουμε, τον, ε, έχουμε την πιο Odgard που είναι υπεύθυνη για την εταιρική υπευθυνότητα του, του, της Ένωσης ε, Δανέζικων Κλώστων Εμφαντουργικών Προϊόντων. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σε αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ε, είναι τιμή μου. Πολύ σύντομη παρουσίαση. Είμαι υπεύθυνη για θέματα κοινωνικής υπευθυνότητας στην ε, οργάνωσή μας που είναι οργάνωση ε, του κλάδου του, της μόδας και των κλωστοφαντουργικών προϊόντων. Εργαζόμαστε για τα θέματα αυτά εδώ και πολλά χρόνια. Τα τελευταία 34 χρόνια κάνουμε καταρτήσεις και μαθήματα για τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για τα θέματα αυτά. Και μπορώ να καταλήξω λέγοντας ότι αν δούμε τις ε, παγκόσμιες κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ, είναι γενικοί κανόνες για τον τρόπο συμπεριφοράς των επιχειρήσεων και από το 2011 έχουμε αυτές τις κατευθύνες γραμμές ε, του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΣΑ. Έχουμε λοιπόν τα αναγκαία μέσα, έχουμε σημεία αναφοράς που τα καλύπτουν όλα. Ήδη περιγράφουν τι πρέπει να κάνουν οι εταιρείε, οι επιχειρήσεις, ποιες είναι οι ευθύνε τους, ποιες είναι οι ευθύνε των πολυεθνικών επιχειρήσεων ποια είναι η ευθύνη των κυβερνήσεων, ποιε είναι οι ευθύνε των διεθνών οργανώσεων. Και επίση τονίζουν ότι μόνο μέσω συνεργασίας και πολυμερών πρωτοβουλειών μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα. Έχουμε λοιπόν τα μέσα, έχουμε το πλαίσιο, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά δεν το κάνουμε. Δεν εφαρμόζονται όλα αυτά ακόμη και υπάρχουν ε, στα κλώστο ή φαντουργικά και στη μόδα μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες οι οποίες είναι τεραστίων διαστάσεων, ε, είναι πολύ μπροστά, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και το κάνουν. Αλλά ας δούμε πώς έχουν τα πράγματα στην ε, Δανία. Περίπου το 59% είναι μικρομεσαίες. Δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τη γνώση, τις δεξιότητες για να συνεργαστούν για αυτό το Παγκόσμιο Σύμφωνο και για να εφαρμόσουν τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Γι' αυτό πριν από τρία χρόνια στο δικό μας ε, οργανισμό για την υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά σχεδιάσαμε κάποια προγράμματα και συζητώντας με τον Υπουργό Ανάπτυξης ε, της Δανίας μας είπε ότι καλή είναι αυτή η προσπάθεια ε, διαμορφώστε ένα πλαίσιο συνεργασίας με τις άλλες οργανώσεις ε, και επιμελητήρια. Πήγαμε στο επιμελητήριο και το Ινστιτούτο του κλάδου μας και αποφασίσαμε ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο εστιάζει σε τρεις τομείς γιατί πρέπει να ασχοληθούμε με διάφορα διαφορετικά θέματα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καλύψουμε το, την έλλειψη γνώσεων και δυνατοτήτων των μικρομεσαίων. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξουν αυτές οι επιχειρήσεις τις δυνατότητές τους για να γνωρίζουν τι μπορούν να κάνουν και ναι, μια μικρή επιχείρηση μπορεί να αναρωτηθεί. Εμείς θα ασχοληθούμε με ανθρώπινα δικαιώματα, δεν έχουμε καμία δυνατότητα. Αλλά υπάρχουν οι καθεντήριες γραμμέ του ΟΗΕ και όλοι πρέπει να το αντιμετωπίσουν με τη δέουσα επιμέλεια. Άρα δεν είναι προσυζήτηση. Ναι, μεν είναι περίπλοκο, αλλά οι οργανώσει του επιχειρηματικού κόσμου πρέπει να τους βοηθήσουν να συμμορφωθούν. Οι τρεις τομείς εστίαση. Πρώτον, να ενισχύσουμε τι δυνατότητες για υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Να ενισχύσουμε τη δυνατότητα για την ε, βελτίωση στις χώρες παραγωγής των συνθήκων ε, εργασίας, των αμοιβών και του περιβάλλοντος. Γιατί όπως ξέρετε το 99% παράγεται εκεί, σε αυτές τις χώρες χαμηλού εργατικού κόστους. Και το τελευταίο, το πολύ σημαντικό, πρέπει να απευθυνθούμε στους καταναλωτές. Πρέπει να μάθουν τι είναι τα βιώσιμα κλώστο υφαντουργικά, να μάθουν οι καταναλωτές ότι αυτά πρέπει να αγοράσουν, να δημιουργήσουμε ζήτηση για αυτά τα βιώσιμα ε, ενδύματα. Οι Δανείοι λένε εμείς δεν παράγουμε τέτοια προϊόντα με αυτή την σημαία, αυτό το έβλημα, το λουλούδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Αλλά πρέπει να το πούμε για να υπάρχει ζήτηση. Πρέπει να το μάθουν οι καταναλωτές, ότι μπορούν να αγοράσουν βιώσιμα ρούχα. Πρέπει λοιπόν το πρώτο είναι να αναπτύξουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Δανία τη δυνατότητα συμμόρφωσης, να ενημερωθούν δηλαδή ότι πρέπει να συνεργαστούν με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με τα συνδικάτα. Δεν μπορούν μόνες τους να αλλάξουν τον κόσμο. Πρέπει να συζητήσουν τα θέματα με τις εταιρείε με τις οποίες συνεργάζονται στις χώρες παραγωγής, γιατί αλλιώς δεν κάνουν το κομμάτι τους της δέουσας επιμέλειας. Μετά πρέπει να πάμε στις χώρες παραγωγής. Και το κάνουμε αυτό ακριβώς με πιο ε, ευέλικτο τρόπο ε, βοηθούμε τις επιχειρήσεις στο διάλογο με τους ε, προμηθευτές τους να φροντίσουν ώστε να τηρούνται οι κανόνες. Και όταν έχουμε λοιπόν τα βιώσιμα προϊόντα τότε πρέπει να τα κάνουμε γνωστά να αυξήσουμε ζήτηση μεταξύ των καταναλωτών για αυτά τα προϊόντα. Στη Δανία. Το πλαίσιο για όλα αυτά είναι οι γραμμές του ΟΣΑ, του ΟΗΕ και κατευθύνει ε, αξίες, αρχές του ΟΗΕ. Μέχρι στιγμή όμως δεν έχουμε λάβει επαρκή χρηματοδότηση για τους δύο τομείς εστίαση, αλλά έχουμε το πρόγραμμα Step Up στο Μαγκλαντές, όπου εργαζόμαστε, και μετά από όλε τις πρωτοβουλίες που ξεκινήσαμε στο Μαγκλαντές, καταλάβαμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τις μεγαλύτερες οργανώσεις των ε, ε, πολιτών. Πήγαμε λοιπόν στην εταιρεία PDMEA στο Μαγκλαντές και τους είπαμε πρέπει να βοηθήσουμε τα μέλη μας για το θέμα αυτό. Αν μπορούμε να συνεργαστούμε μαζί σας, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς τα θέματα εδώ επιτόπου. Και για ποιο λόγο. Όχι για να τους δημιουργήσουμε δυνατότητες, για να καταλάβουν όλοι ότι έχει έννοια και η οικονομική, η σωστή κοινωνική συμπεριφορά. Η συμπεριφορά ε, με κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τις εταιρείες εκεί, λοιπόν, και είμαστε τώρα σε φάση όπου συνδυάζουμε την κοινωνική υπευθυνότητα με βελτίωση και των προϊόντων. Γιατί η Μαγκλαντές θέλει να βελτιωθεί η παραγωγικότητα. Διότι είναι κακή εικόνα του στον τύπο. Προσπαθούμε λοιπόν να προωθήσουμε, να αυξήσουμε και την παραγωγικότητα για να, κερδιθεί, ε, για να υπάρξουν κέρδη τα οποία να δαπανηθούν σε υπευθυνότητα. Πρόεδρος. Είναι σαφέ το μήνυμα, έχουμε δυνατότητα, ά το κάνουμε. Και τώρα, ο Γιώργο Αλτιντζή. Υπεύθυνο οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής από τη Διεθνή Συνομοσπονδία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Ευχαριστώ πολύ, Στέλιο. Θα αρχίσω λέγοντας ότι οι παγκόσμιες αλυσίδες ε, αξιών είναι ένα μέσο για την ανάπτυξη σε γενικές γραμμές. Υπάρχουν ωστόσο πολύ σοβαρά προβλήματα και σημαντικές ελλείψεις, οι οποίες έχουν εντοπιστεί στα αποτελέσματα του συνεδρίου του, της Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας. Σε εντοπίστηκαν μάλιστα από όλους τους φορείς. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν κυρίως για δύο λόγους. Από την αρχή, ε, αρχικά, από αυτόν τον αγώνα προς την κατώτερη τιμή και από σοβαρές ασυμμετρίες και ανισορροπίες που υπάρχουν μέσα στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού. Δηλαδή, οι μεγάλοι αγοραστές έχουν πολύ δύναμη, έχουν πολλούς παραγωγούς Γι' αυτό λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι στις κατώτερες βαθμίδες της ε, παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού, είναι πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες ε, αξιοποίησης αυτής της αξίας. Έχω κάποιες διαφάνειες μαζί μου που περιλαμβάνουν μια ανάλυση το πόσο κοστίζουν αυτά τα τζιν των 22 δολαρίων, το πώς δηλαδή διανέμεται αυτή η αξία στους διάφορους ε, τομείς. Το εργοστάσιο λοιπόν στον Μπαγκλαντές βγάζει 1,16 δολάρια από τα 22, από τα οποία 1,16 δολάρια 90 cents είναι το κόστος του εργοστασίου, είναι και το κέρδος αυτής της μικρής επιχείρησης και μόνο 26 cents πηγαίνουν στους εργάτες του εργοστασίου. Κάτω δηλαδή από το 1% του κέρδου πηγαίνει στου ε, εργάτες και πολλές φορές αυτό το ποσοστό φτάνει το 0,6%. Μετά, διανομής, ε, μεταφορής τα καταστήματα, όλες οι άλλες ε, επόμενες διαδικασίες καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας αυτή την αλυσίδα αξιών. Ο, ε, ο Γενικός Διευθυντής του, της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας έγραψε ότι το έγγραφο της οργάνωσης το, ε, δίνει έμφαση στους τρόπους με τους οποίους ορισμένες ε, επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτές τις δυσμενείς επιπτώσεις. Δηλαδή, η ανάκληση λάθος αποφάσεων, οι οποίες αφορούν μείωση κόστους μέσω της μείωσης των εργασιακών της επιδείνωσης των εργασιακών συνθήκων. Τι εννοούμε εδώ, ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες όπου ε, ιδρεύουν οι περισσότεροι προμηθευτές δεν έχουν επαρκή νομοθεσία ή εάν έχουν δεν εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία ε, επαρκώς. Έτσι δημιουργούνται αυτά τα κενά και μετά δημιουργείται ένα περιβάλλον ευνοϊκό προς ε, αυτές ε, τις ε, άσχημες επιχειρηματικές πρακτικές. Δηλαδή, χρησιμοποιούν και εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το γεγονός ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν ορισμένες χώρες την νομοθεσία τους. Και στην περίπτωση του Μπαγκλαντές έχουμε το εξής. Ακούσαμε τον Υπουργό Εργασίας να λέει ότι θεωρεί τη φτηνή εργασία ένα από τα πλεονεκτήματα που κάνουν ανταγωνιστική τη χώρα του. Είναι λοιπόν μια εσκεμμένη πολιτική να ε, καταστέλλονται τα συνδικάτα και να ε, είναι η μισθή όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Αυτό φυσικά έχει οδηγήσει σε ημερομίσθια τα οποία είναι κάτω από το κατώτατο όριο, δεν επαρκούν για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Πολλοί εργάζονται ε, από το σπίτι, πολλοί είναι γυναίκες και εργάζονται σε συνθήκες που λίγο διαφέρουν από συνθήκες δουλείας. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις τα πράγματα είναι έτσι στις αναπτυσσόμενες χώρες. Τώρα, πέρασα δύο εβδομάδες. Ε, εκεί είχαμε εκτενείς ε, συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με εκπροσώπους των εργοδοτών με χαρά μου διαπίστωσα ότι πολλές κυβερνήσεις και εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στήριξαν το σκοπό για τον οποίο αγωνιζόμαστε. Οι αποφάσεις της ε, Διεθνής Οργάνωσης Εργασίας μετά από το συνέδριο αναφέρουν ότι χρειάζεται οι κυβερνήσεις να προωθήσουν τον ενεργό κοινωνικό διάλογο. Εδώ αναφέρθηκαν σε παγκόσμιες συμφωνίες πλαίσιο με μεγάλες εταιρείε και μεγάλες συνομοσπονδίες που χρειάζεται να υπογράψουν συλλογικέ συμβάσει. Επίση, χρήση των δημόσιων συμβάσεων για να προωθήσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα σε, όλο, σε όλα τα στάδια της ε, αλυσίδα εφοδιασμού. Πρόταση να αρχίσει η διαδικασία της δέουσας επιμέλειας πρώτα στις δημόσιε δημόσιες επιχειρήσεις, στις κρατικές επιχειρήσεις μάλλον, και Υπάρχει η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ευνορικό περιβάλλον που θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν διαδικασίες δέουσας επιμέλειας στην διοίκησή τους. Στην επόμενη πρόταση ε, αναφέρεται τι χρειάζεται η πλευρά της διακυβέρνησης να ε, ζητήσει από τις επιχειρήσεις. Τι χρειάζεται να γίνει νομοθετικά. Αυτό το τελευταίο έγγραφο περιλαμβάνει μια πρόταση να γίνει μια αξιολόγηση της κατάστασης το ερχόμενο έτος, η οποία ενδεχομένως οδηγήσει σε μια σύμβαση. Εκεί αυτό που ζητούμε εδώ και χρόνια είναι η δέουσα επιμέλεια να γίνει υποχρεωτική. υποχρεωτική απέτηση για όλες τις επιχειρήσεις. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και κάποιες συνέπειες. Και πρέπει να παρέχονται τα σωστά μέσα αντιμετώπισης καταχρήσεων. Ωστόσο, θα ανάγκαζα ένα τέτοιο υποχρεωτικό χαρακτήρα να αλλάξουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο οι μεγάλες πολυεθνικές που είναι υπεύθυνε, Δηλαδή θα γίνει εσωτερήκευση του εξωτερικού κόστους έτσι ώστε να φαίνεται με περισσότερη σαφήνεια ε, το τι γίνεται, το ποια στάδια ακολουθούν. Τώρα, ε, η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας και όσα θα πρέπει να αποκρισταλώσουν αυτή τη δέουσα επιμέλεια, να δώσουν έναν ορισμό έτσι ώστε να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μας δώσατε μια διαφορετική απόχρωση της κατάστασης. Τώρα θα αρχίσει ο κύκλος των ερωταπαντήσεων. Άρνε Λίτς, έχετε το λόγο. Πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις διαφορετικές οπτικές γωνίες που μας δώσατε. Πολλοί από εσά μου είστε γνώριμοι, διότι τα τελευταία δύο χρόνια ε, με απασχολεί το θέμα της ε, κλωσοφαντουργία και της ένδυσης. Χαίρομαι πολύ που έχει έρθει εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έχει αναλάβει τα ενία σε αυτή την πολύ δύσκολη προσπάθεια να κάνει αυτή την ανάλυση. Πολλές ε, διευθύνσεις της Επιτροπής συνεργάζονται για αυτό το κείμενο και θεωρώ πολύ σημαντικό το ότι έχουμε αυτό το κείμενο. Είναι μια αφετηρία η οποία θα προσπαθήσει να φέρει τα πράγματα πιο πέρα. Επίσης, άκουσα και την παρέμβαση από τη Δανία με μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρατε, δεν θυμάμαι ποιος, νομίζω ανέφερε πρόσωπος της ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου, ότι παίζουν μεγάλο ρόλο και οι εθνικές πρωτοβουλίες. και αναμένοντας τα τελικά αποτελέσματα της έρευνα του τι ακριβώ συμβαίνει την Ευρώπη, βλέπω ότι η πρωτοβουλία της ε, Δανία είναι ένα τέτοιο παράδειγμα εθνικής ε, πρωτοβουλίας. Νομίζω και όλες ότι η Γαλλία, οι κάτω χώρες και η Γερμανία έχουν μεγάλο δυναμικό εδώ. Η Γαλλική Προεδρία μάλιστα επέμεινε σε αυτό. Και χαίρομαι πάρα πολύ ε, για το ότι μέχρι τις 4 Ιουλίου η Ολλανδική Προεδρία θα υποβάλει μία πρόταση για ε, τα εφάσματα και για την φαντουργία. και χαίρομαι πάρα πολύ που ε, υπάρχει εδώ και εκπρόσωπος από τα συνδικάτα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω τι πρωτοβουλίες υπάρχουν και ποιες θεωρείτε πως είναι αρκετά προοδευτικές και τι μελιγενέστε εκεί. Αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν 7 εθνικές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη. Βλέπω λοιπόν ότι αυξάνεται το δυναμικό και οφείλεται αυτό στις προσπάθειες του κύριου Μίμητσα φαντάζομαι. Τώρα από την πλευρά και των επιχειρήσεων αλλά και των εργαζομένων, ποιο θεωρείτε εσείς ότι είναι ένα καλό ε, επιχειρησιακό μοντέλο και Ελπίζετε να καταλήξουν όλες αυτές οι προσπάθειες σε ένα ψήφισμα, το οποίο δεν θα αφορά μόνο την ανάπτυξη, αλλά κυρίως και το εμπόριο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρείτε πως η Ολλανδική Προεδρία έχει κάνει καλή δουλειά και πώς θα έπρεπε να μεταβούμε στην επόμενη Προεδρία, πώς θα έπρεπε να ε, γίνει μια ομαλή μετάβαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους ε, εισηγητές ε, για την εισαγωγή τους. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε πως ένα από τα πιο καυτά θέματα είναι πως θα μπορέσουμε να οργανώσουμε μια ε, αλυσίδα αξίας που θα λαμβάνει υπόψη και τον περιβαλλοντικό και τον ανθρώπινο παράγοντα. Και Προφανώς όλοι συμφωνούμε με όλα όσα είπατε για την κατάσταση στον Μπαλκλαντές. Και επίσης ο πρόεδρος μίλησε και για το θέμα του τριμερούς διαλόγου που έχουμε σήμερα το απόγευμα και όλων των ε, αντιπαραθέσεων. Ε, ε, προσπαθούμε να έχουμε όσο και όλο και περισσότερο υποχρεωτικές ρυθμίσεις για την συνεργασία και στην εφοδιάζουσα βιομηχανία και στην ε, βιομηχανία που βρίσκεται στην άλλη πλευρά της αλυσίδας. Όμως, είναι και θέμα πολιτικής βούλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες. Να υπάρξει δηλαδή ένα τέτοιο πλαίσιο συνεργασίας που θα πλαισιώνει την συμφωνία, την προσέγγισή μας και θα οργανώσει το εμπόριο στο επίπεδο της παραγωγής αλλά και της κατανάλωσης. Μπορούμε να βρούμε την συγκεκριμένη απάντηση στην κατάσταση που παρουσιάσατε μόνο αν παρουσιάσουμε συγκεκριμένες λύσεις στο τραπέζι. Ίσως εσείς να έχετε κάποιες απαντήσεις λοιπόν για το ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό διαβούλευσης για να παρακολουθούμε τη διαφθορά της κυβέρνησης και την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις ικανότητες που έχουμε να πείσουμε τους νομοθέτες. Ναι, ναι, θα τελειώσω. Με ποιον τρόπο χρησιμοποιούμε τις υφιστάμενες καθευθυντήριες γραμμές του ΩΣΑ για να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμες αξίες. Μιλήσατε για τη δημιουργία των τιμών, εξωτερικοποίηση των τιμών για να κάνουμε μια εσωτερικοποίηση. Πώς θα συνδυάσουμε το δικό μας έργο με την Επιτροπή ΙΜΠΟ, με την Επιτροπή ΙΝΤΡΕ, έτσι ώστε να έχουμε διαμορφώσει και τους κανονισμούς της εσωτερικής αγοράς. Αυτή είναι η πρόκληση που όλοι μας αντιμετωπίζουμε, να είμαστε πιο υπεύθυνοι, πιο ακριβείς στη δουλειά μας, ο καθένας στον τομέα του. Κύριε ναι. Ε, το ερώτημα είναι πώς διασφαλίζουμε ότι οι αλυσίδες αξίας είναι βιώσιμες με όλους τους τρόπους που αναφέραμε. Νομίζω ότι υπάρχουν κάποια όρια στην δέουσα επιμέλουσα, επιμέλεια. Ε, προωθούμε και θα προωθήσουμε. Οπότε αυτό όμως δεν φτάνει. Και θέλω να ακούσω τη δική σας άποψη γι' αυτό το να επικεντρωθούμε απλώς στις εκθέσεις σχετικά με το τι έχει γίνει ως τώρα, ε, ίσως είναι λίγο. Ε, θέλουμε να δούμε τι θα γίνει ε, αν κάτι πάει στραβά, γιατί προς το παρόν οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες. Εμείς ως νομοθέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι απλώς δεν παρακολουθούμε και δεν κάνουμε εκθέσεις όταν ε, κάτι πάει στραβά και πώς θα μπορέσουμε να σταματήσουμε ε, τα προβλήματα. Τελευταία η, η, Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ε, ομιλητές για τη συμμετοχή τους σε αυτή την ακρόαση και θέλω να κάνω μια ερώτηση. Στο περιθώριο όλων όσα είναι αναγκαία να κάνουμε για να βελτιώσουμε τους κανόνες της παγκοσμιοποίηση και ιδιαίτερα των αλυσίδων αξία, αυτό που θα είναι πολύ δύσκολο, όπω είπε και ο εκπρόσωπο των συνδικάτων, και να είναι υποχρεωτική ιδέουσα επιμέλεια, αυτό πρέπει να το επιδιώξουμε. Παράλληλα, θα ήθελα να μου πείτε πώ μπορούμε μέσω των δημοσίων συμβολέων να απαιτούμε ότι οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση είτε μέσω απευθείας συμβολέων είτε μέσω υπεργολαβιών θα πρέπει να εκτελούν αυτή την δέουσα επιμέλεια γιατί πρέπει να αποκτήσουν κοινωνική υπευθυνότητα οι επιχειρήσεις πρέπει να αλλάξουν οτροπή να καταλάβουν ότι όλοι είναι υπεύθυνοι για τη σωστή αυτή στάση. Επίσης, τι ακριβώς περιμένετε, τι περισσότερα περιμένετε ότι θα μπορούσε να κάνει το Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να επιτύχουμε την καλύτερη εφαρμογή και καλύτερους κανόνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Εμμανουέλ Μπουτόν Στάμπς. Είναι η συντάκτρια γνωμοδότησης της ε, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής για ε, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. GVC. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε, Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση ε, είναι διαθέσιμη στην είσοδο εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα, μόνο μία ψήφος κατά ε, τον Μάιο. Υπήρχε πολύ καλή συνεργασία όλων των πολιτικών ομάδων στην ΟΚΕ μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων. Το θέμα είναι περίπλοκο όπως υπόθηκε. Η προσέγγισή μας ήταν να βασιστούμε σε στοιχεία, να περιγράψουμε τη λειτουργία ορισμένων τέτοιων ε, αλυσίδων και εξετάσαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις ε, ηλεκτρονικός κλάδος και ένδυση. Πολύ ενδιαφέρουσες αλυσίδες γιατί ο ρόλος των υπεργολάβων, ο ρόλος των ε, προμηθευτών είναι πολύ διαφορετικός και πολύ διαφορετικές και οι κοινωνικές προκλήσεις για την ένδυση όπως ήδη υπόθηκε είναι ότι η μισθή δεν είναι βιώσιμη, καταναγκαστική εργασία, παιδική εργασία, αλλά για ηλεκτρονικά προϊόντα είναι διαφορετικά τα προβλήματα. Μερική απασχόληση, ε, υπερβολικές ώρες εργασίας, πρόσβαση στην κατάρτιση. Πολύ διαφορετικά. Και επίσης ε, περιγράφουμε και πολλές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει σε διάφορα επίπεδα, διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, από πλευράς διεθνών οργανώσεων και είναι πολύ ενδιαφέρον να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει καλή συνεργασία δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και υπάρχει ακόμη πολύ περιθώριο για να γίνουν πιο γνωστές οι βέλτιστες πρακτικές. Η γνωμοδότησή μας ε, είναι μόλις 8 σελίδες, περιέχει πολλές από τις συστάσεις. Πολλές συστάσεις ε, και να αναφέρω μερικές. Το πρώτο είναι να υπάρξει μια σωστή διευκρίνηση για το τι ρόλο παίζει ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας. Δεν μπορεί να ζητήσει κανείς από μια πολυεθνική να κάνει τη δουλειά μιας κυβέρνησης. Και δεν μπορούμε να ζητήσουμε από ένα Δήμο που πολύ συχνά δεν έχει επαρκείς πόρους να είναι τόσο ισχυρός όσο μια πολυεθνική. Πρώτα λοιπόν πρέπει να διευκρινιστεί ο ρόλος του κάθε εμπλεκομένου. Δεύτερον, πρέπει να μάθουμε περισσότερα για το πώς λειτουργούν τώρα αυτές οι αλυσίδες. Χρειαζόμαστε περισσότερα στατιστικά στοιχεία, χρειαζόμαστε καλύτερη χρήση των βάσεων δεδομένων του ΠΟΕ για τις αλυσίδες και επίσης πρέπει να πιέσουμε ούτω ώστε να υπάρξει ένα πολύ φιλόδοξο αλλά και πολύ συνεπές και ολοκληρωμένο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει μια ενιαία πολιτική και εντός και εκτός. Και για την εσωτερική αγορά πρέπει να κάνουμε πολλά για τις δημόσιες προμήθειες, για την σήμανση για παράδειγμα, γιατί πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Διαφάνεια και έναντι του τελικού καταναλωτή. Πρέπει επίσης να ευνοήσουμε και να γνωστοποιήσουμε τις πολλές καλές πρακτικές θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε, για παράδειγμα, τη μορφή μιας ε, συμμαχίας ε, πολλαπλών εμπλεκομένων. Είναι πιο κατάλληλη μορφή. Και επίσης, στηρίζουμε και διάφορες πρωτοβουλίες επιτόπου με πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέσα για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν ε, την κατανόηση των για το ποιες προκλήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν. Για παράδειγμα, δυνατότητες αυτοαξιολόγησης. Και όπως λέει και η δήλωση του ε, Διεθνούς Οργανισμού ε, Εργασίας, πρέπει να υπάρξει κοινωνικός διάλογος, πολύ πιο ευρύτερος ε, για καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και από πλευράς εργαζομένων και από πλευράς εργοδοτών. Σας ευχαριστώ και εγώ που ήρθατε και μας παρουσιάσατε τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕΜ. Πρωτού τώρα δώσω το λόγο στους εμπειρογνώμονες. Δύο λεπτά έχει ο καθένας σας για να αντιδράσει στα σχόλια και τις ερωτήσεις. Θα κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Δεν μας ικανοποιεί η στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρωτοβουλία για ε, την ένδυση. Εδώ και πολύ καιρό περιμένουμε κάποια πρόταση. Και μάλιστα στα αυτήν εδώ την αίθουσα πριν από λίγες εβδομάδες είχαμε έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν ήταν και τόσο ευχάριστα αυτά που ακούσαμε. Ακόμα λοιπόν και αν δεν θα μας κάνετε κανένα δώρο για τα Χριστούγεννα θα μπορούσατε ίσως να λάβετε υπόψη την επιθυμία του Κοινοβουλίου να αναλάβετε δράση για την ένδυση και την κλωστοεφαντουργία. Τώρα θα αρχίσω αντίστροφα, θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο της Διεθνής των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Μόνο δύο λεπτά έχω. Αν είχα δύο ώρες καλύτερα θα ήταν. Τώρα, ποιες εθνικές πρωτοβουλίες είναι οι καλύτερες, νομίζω, με ρώτησαν αρχικά. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχουμε υποστηρίξει επίσημα κάποια πρωτοβουλία δεν έχουμε χαρακτηρίσει κάποια ω καλύτερη. Υπάρχουν όμως πολλές που έχουν καλά στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία που έχουμε εντοπίσει ως αναγκαία στις εθνικές πρωτοβουλίες είναι τα εξή δύο. Ε, συμβάσεις ανάμεσα στην κεντρική, ε, στην μεγάλη ε, εταιρεία και στις μικρότερες πρέπει να γίνουν άμεσα, όσο το δυνατόν περισσότερο, από έμεσα άμεσα. Δεύτερον, βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, συμβάσεις να γίνουν μακροπρόθεσμες. Δηλαδή, όταν μια μικρή επιχείρηση, ε, πολύ πιο μετά στην αλυσίδα, έχει μια άμεση σύμβαση κατευθείαν με την μεγάλη την κεντρική εταιρεία, τότε θα έχουν πολύ καλύτερες δυνατότητες ε, αντιμετώπισης των εργαζομένων τους, καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας. Μετά, κάτι άλλο πρόθεση, ενεργός πρόθεση των συλλογικών εμπορικών συμβάσεων. Όπως είπα και πριν υπάρχουν συμφωνίες με ε, διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και ε, επιχειρήσεις από τη μία και από την άλλη πρέπει να προωθηθούν τα συνδικάτα. Κανένας δεν είναι καλύτερος επιθεωρητής από ένα συνδικάτο. Αυτό ε, βοηθά και σε χώρες τις οποίες δεν υπάρχουν επιθεωρητές εργασίας. Θα θέλαμε εδώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της. Τώρα, στην ομάδα των εργαζομένων στην Παγκόσμια Οργάνωση Εργασία ε, επιχειρηματολογούμε ότι δεν έχουν οδηγήσει όλες τις πρωτοβουλίες τα καλά αποτελέσματα. Ξέρουμε πώς μπορεί να υπάρχουν καλές προθέσεις από τους ε, εργοδότες και από τις επιχειρήσεις και αυτές ε, πρέπει να είναι οι πρωτοβουλίε που θα εστιάσουμε. Τώρα, στο συνέδριο συζητήθηκε επίσης και η προστασία όσων καταγγέλουν παρατυπίες. Αυτό έχει επαναληφθεί σε πολλές ε, περιπτώσεις. Σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αναφοράς ε, καταγγελιών και πρέπει να υπάρχει και ιδέουσα επιμέλεια όπου θα εξετάζεται περισσότερο ε, αυτή η καταγγελία. Τώρα, άλλη ερώτηση, τρίτη ερώτηση. Ποια μέσα διαθέτουμε. Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί αποζημίωσης που συμφωνούν και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει ο ρόλος των συνδικάτων. Πέρυσι, η καγκελάριος Μέρκελ ε, μίλησε για το ε, Ταμείο Vision Zero, το οποίο είναι ένα ταμείο που αποζημιώνει τους εργάτες σε περίπτωση ατυχήματος. Και ασφάλιση. Πρέπει να εξασφαλιστεί οι ασφαλιστικές εταιρείες σε περίπτωση ατυχήματος να πιέσουν την κορυφή της αλυσίδας, την πηγή του προβλήματος για να αλλάξει το σκηνικό. Και πολύ σύντομα να πω δύο άλλα πράγματα. Ε, δημόσιες προμήθειες. Υπάρχουν πολλές κυβερνήσεις που χρησιμοποιούν κοινωνικές ρήτρε. Γιατί λοιπόν να μην χρησιμοποιούν και την αρχή της δέουσας επιμέλειας. Δυστυχώς, ε, το έγγραφο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας δεν ε, γίνεται λόγος γι' αυτό. Τώρα, εσείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ήταν ε, ιδανικό εάν μέσα σε ένα κείμενο ζητούσατε να γίνει υποχρεωτική ιδέουσα επιμέλεια, ίσως αρχίζοντας σε πιο ήπια, με εξοδευτική ευθύνη και προχωρώντας στη συνέχεια. Επίσης, πρέπει να αναπτυχθούν δυνατότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ενισχυθούν τα συνδικάτα και οι ενώσεις εργαζομένων και ίσως αυτές οι συζητήσεις να οδηγήσουν του χρόνου σε κάποιο συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ. Η Πία έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Όσον αφορά στο πρώτο ερώτημα που αναφέρατε, τις διάφορες πρωτοβουλίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν ε, ολοκληρωμένες πρωτοβουλίες και πολύ καλές στην ε, Γερμανία και την Ολλανδία που είναι ηγέτης. Συνεργαζόμαστε και με τη Γερμανία και με την Ολλανδία και θα θέλαμε να συνεργαστούμε και με άλλους, αλλά όπως είπε και ένας άλλος ομιλητής, κάτι πολύ έξυπνο, πρέπει να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πρέπει αυτός ο νέος τρόπος εργασίας βάσει της δέουσας επιμέλειας να εξερευνηθεί, να το μάθουμε πριν ε, αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις άλλες χώρες, να έχουμε εμπειρία πριν πούμε ότι αυτό λειτουργεί για μας, ε, να δούμε πώς λειτουργεί και για σας, να δούμε πώς θα συνεργαστούμε για να αποκρισταλώσουμε την καλύτερη λύση. Τώρα για την ε, υποχρεωτική ιδέουσα επιμέλεια να αναφερθώ σε μία αξιολόγηση που έχει κάνει η επιχειρηματική αρχή της Δανίας για διάφορα ζητήματα ένα από αυτά είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη και αξιολόγησαν τι ακριβώς είναι αυτό που θα φέρει τα καλύτερα ε, αποτελέσματα. Κάτι υποχρεωτικό, ένας κανονισμός ή μια ε, εθελούσια προσέγγιση. Φαίνεται λοιπόν ότι η ε, Θελούσε συμμετοχή δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα γιατί στις υποχρεωτικές ε, ε, προσεγγίσεις απλώς τσεκάρεις τα κουτάκια και λες αυτό το έκανα και αυτό το έκανα. Εμείς θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Θέλουμε οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης να ενσωματωθούν και στις επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε απλώς να τσεκάρουμε του κουτάκια. Θέλουμε να έχουμε μια ευρύτερη άποψη για το τι χρειάζεται να γίνει και να περιλάβουμε και ε, τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι ε, η εθελοντική συμμετοχή έχει καλύτερα αποτελέσματα γιατί αναλαμβάνεις την ευθύνη, ε, θέλεις να κάνεις τη δουλειά και την κάνεις. Αν είσαι υποχρεωμένος, το κάνεις μόνο και μόνο για να πεις ότι το έκανες. Θέλουμε λοιπόν να προωθήσουμε την εθελούσια προσέγγιση και σε μερικά χρόνια από τώρα να εξετάσουμε αν λειτουργήσε. Δεν μας ενδιαφέρει λοιπόν να έχουμε περισσότερη νομοθεσία στο θέμα της δέουσας επιμέλειας. Νομίζω ότι τα Ηνωμένα Έθνη έκαναν πολύ καλή δουλειά. Έχουν καθορίσει ξεκάθαρα ποια είναι η δουλειά των επιχειρήσεων και ποια των κυβερνήσεων και πώς μπορούν να συνεργαστούν και να συμπεριλάβουν και άλλους ενδιαφερόμενους για να επιτευχθούν οι στόχοι. Αυτά ήθελα να πω για αυτό το θέμα και να απαντήσω τώρα στην ερώτηση για το θέμα του πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα και να μην κάνουμε απλώς εκθέσεις. Αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε μια διαδικασία δέουσας επιμέλειας και να ακολουθήσουμε όλα τα στάδια, δεν έχουμε απλώς ε, κάτι που γίνεται τυπικά. Πρέπει να βουτήξουμε πιο βαθιά. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Τσέρι. Κυρία Σέρι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, ε, από η οποία κυρίως ε, είχε να κάνει με τον τρόπο συμπεριφοράς ε, των εταιριών και το πώς οι κυβερνήσεις επηρεάζουν αυτή τη συμπεριφορά. Εγώ να σας πάω δύο επίπεδα πάνω για να μπορέσω να βγάλω τα συμπεράσματα βάσει των όσων είπα στην ομιλία μου για το Διεθνές Σύστημα Εμπορίου. Να επιστήσω λοιπόν την ε, προσοχή σας στις, ε, στα συμπαράσματα του ICTST και του Παγκόσμιου Οικονομικού ε, φόρουμ για την περίοδο 2012-2015, όπου υπήρχαν ομάδες εμπειρογνωμόνων, μία για τις ε, αλυσίδες αξίας και έδωσαν συστάσεις σχετικά με το τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση. Και μπορείτε να δείτε τη σχετική έκθεση. Ε, υπάρχει το link στα έγγραφα που δόθηκαν για αυτή τη συνεδρίαση. Κάποιες λοιπόν από τις επιλογές που υπάρχουν ε, ε, είναι η εξής, η ανάπτυξη και βελτίωση των εργαλείων γνώσης για να έχουμε μια πιο εμπειρική και λεπτομερή κατανόηση των, αξιών, των αλυσιδών αξίας. Είναι βάση ε, των συστάσεων του ΕΕ. Ηνωμένων Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ανεξάρτητη πλατφόρμα η οποία θα εξετάζει πώς λειτουργούν οι αλυσίδες αξίες ε, για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Ποιες είναι οι, αξίες, οι αλυσίδες που τις ε, ωφελούν περισσότερο. Πώς ε, γίνεται ανταλλαγή, πώς μπορεί κανείς να πάει πέρα από τις αλυσίδες αξίας. Όλα αυτά δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί. Και αυτό πάλι αναφέρεται στη σύσταση του ECOSOC. Τέλος, να σκεφτούμε πώς θα ε, διερευνήσουμε την ανάγκη για νέα διεθνή πλαίσια, για βασικές πολιτικές που θα επηρεάσουν ε, τη λειτουργία. Μπορεί να έχουμε πολυμερείς πρωτοβουλίες για την επένδυση, το ανταγωνισμό, την, ε, το ψηφιακό εμπόριο. Όλα αυτά θα υποστηρίξουν τις τρέχουσες δραστηριότητες και αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να τα υπερασπιστεί μέσω των πρωτοβουλειών της για το εμπόριο. Ωραία. Σχεδόν τελειώνουμε. Υπήρξαν πολλές καλές προτάσεις και συστάσεις. Ήταν πολύ επικοδομητική η συζήτηση νομίζω. Ο κύριος Πρόεδρος της Επιτροπής ΙΝΤΑ θα συμφωνεί μαζί μου ότι πρέπει να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Εκ μέρους της Επιτροπής λοιπόν Ανάπτυξης, ευχαριστώ πολύ τους ομιλητές, τους συναδέλφους για όλη τη συζήτηση. Θα επανέλθουμε, σωστά. Ευχαριστώ. Φυσικά θα επανέλθουμε αφού συνεργαζόμεθα για τα κλωστοεφαντουργικά αλλά και για άλλα. Καλή συνεργασία είχαμε και για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων. Σας ευχαριστώ που συμπροεδρεύσαμε και τώρα έχουμε το δεύτερο γύρο ομιλιών που θα ασχοληθεί με τα γεωργικά. Πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα και εδώ. Πρώτα έχουμε την Κοαλή Νταβίντ από τον ΟΣΑ. Είναι υπεύθυνη του προγράμματος για επενδύσεις στη Γεωργία. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω τι κάνει ο ΟΣΑ για να προωθήσει την υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων στον γεωργικό και τροφιμικό τομέα. Θα ασχοληθώ με πρόσφατες εξελίξεις στο νομοθετικό και πολιτικό τομέα πριν σας περιγράψω τις κατευθύνες γραμμές του ΩΣΑ και πώς βοηθάμε την εφαρμογή τους. Λοιπόν, εδώ είναι τα βασικά πρόσφατα ε, γεγονότα, οι δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι χώρες του ΩΣΑ, η τελευταία υπουργική συνάντηση το 2015 κάλεσε τον ΩΣΑ να συνεχίσει τις προσπάθειες να διευρύνει την, συμμόρφωση, την ε, λειτουργία των Εθνικών Σημείων Επαφής NCP τον Ιούνιο του 2015 οι ηγέτες του G7 κατέστησαν σαφές ότι η υπεύθυνη εταιρική συμπεριφορά ήταν κύρια προτεραιότητα και θέλησαν να εφαρμοστούν καλύτερα τα διεθνή πρότυπα και ενθαρρύνουν τις εταιρείες να εφαρμόσουν την δέουσα επιμέλεια. Τον Δεκέμβριο του 2015 στο Άμστερνταμ έγινε μία δήλωση από πέντε χώρες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, απερίμωση και πρόσφατα τον Απρίλιο ενθαρρύνουν οι Υπουργοί Γεωργίας ε, να ακολουθούν οι υπεύθυνες ε, συγγνώμη, κατευθύντες γραμμές του ΟΣΑ και του ΦΑΟ για υπεύθυνη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Ποιε είναι οι τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις. Έχουμε την οδηγία του 14 της Ένωσης. Πέρυσι, το Μάρτιο λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο πέρασε το νόμο για την σύγχρονη δουλεία που υποχρεώνει τις ε, μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν μια αιτήσια δήλωση για τη δουλεία και τη διακίνηση ατόμων και να κάνουν έκθεση για την δέωση επιμέλεια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπήρχε ένα κενό το οποίο έκλεισε στο νόμο για την επιβολή του εμπορίου και τη διευκόλυνση του εμπορίου έκλεισε τον προηγούμενο Μάρτιο απαγορεύει την εισαγωγή προϊόντων που παράγονται μέσω καταναγκαστικής εργασίας. Και στη Γαλλία ε, είναι που εξέτασε ένα νομοσχέδιο που θα υποχρέωνε τις μεγάλες γαλλικές εταιρείες να αναφέρονται για τη δέωση επιμέλεια στην αλυσίδα τροφοδοσίας τους. Ποιε είναι τώρα οι γραμμές του ΟΣΑ για τις πολυεθνικές. Και μετά θα σας πω τι κάνουμε στον αγροτροφημικό κλάδο. Οι κατευθύνες γραμμές είναι το πιο εκτεταμένο μέσο για τον τομέα αυτό και αφορούν τις πολυεθνικές που εργάζονται σε ή από τις χώρες ε, του ΟΣΑ της 35 αλλά και άλλες 11, συνολικά 46. Οι, οι άλλες είναι στην Λατινική Αμερική και την Αφρική. Εγκρίθηκε πριν από 40 χρόνια, αλλά ενημερώνεται τακτικά η τελευταία ενημέρωση. Εισήγαγε νέα μέτρα για τη δέουσα επιμέλεια. Και αυτοί, αυτές οι κατευθύντριες γραμμές περιέχουν ένα μηχανισμό εφαρμογής που λέγεται ακριβώς εθνικά σημεία επαφής. Σε κάθε χώρα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο σημείο επαφής στα πλαίσια των υπηρεσιών της χώρας. Μπορεί να είναι σε ένα Υπουργείο, μπορεί να είναι τριμερές με τις οργανώσεις των ε, επιχειρήσεων και την κοινωνία των πολιτών πρέπει να προωθήσει τις καθευθυντήριες γραμμές αλλά να ασχοληθεί και με την επίλυση προβλημάτων. Όταν μια οργάνωση, για παράδειγμα, της κοινωνίας των πολιτών θέτει κάποιο ζήτημα, ότι δηλαδή κάποια επιχείρηση δεν τηρεί τις κατευθυντήριες γραμμές. Από το 2000 έχουν ε, υποβληθεί 360 θέματα σε αυτά τα NCP. Βλέπετε ανατομέα και ανακλάδο μάλλον και ανατομέα ποια είναι η κατανομή. Ε, πρόσφατα είχαμε πολλές υποθέσεις για τον γεωργικό τομέα και τον τομέα των τροφίμων, πολύ συγκεκριμένα. Έχουμε το φινικέλαιο στην Ινδονησία. Ήταν ε, μία προσφυγή των φίλων ε, της γης στην Ολλανδία, στο NCP στην Ολλανδία. Και είχε να κάνει με τη δέουσα επιμέλεια. Υπήρξε μία διαδικασία διατησίας, μετά την οποία η Rabobank, που ήταν η επιχείρηση που εμπλεκόταν, συμφώνησε να συνεχιστεί ο διάλογος με όλους τους ενδιαφερομένους εφόσον υπήρχαν ε, στοιχεία ότι η πολιτική της για το Φινικέλο δεν εφαρμοζόταν σωστά και συμφώνησε να τροποποιήσει την αντιμετώπιση προσφυγών. Τη διαδικασία αντιμετώπισης προσφυγών νομίζω ότι απεδείχθη έτσι η χρησιμότητα των ε, σημείων επαφής αυτών ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να εφαρμόζουν τη δέουσα επιμέλεια. Τώρα στον τομέα γεωργίας και τροφίμων για να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις καταλήξαμε στην ε, βοήθεια προς τις επιχειρήσεις μέσω ε, προτάσεων ΟΣΑ και ΦΑΟ. Συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. Ε, δύο έτη κράτησε η διαδικασία καθορισμού αυτού του κειμένου. Θέλουμε να υπάρξει συγκεκριμένη πολιτική αλλά και διαδικασία για σεβασμό αυτής της σωστής πολιτικής των επιχειρήσεων. Ποια είναι αυτή η σωστή, το πρότυπο πολιτικής. Βλέπετε όλα τα είδη των ε, κινδύνων που καλύπτουμε, των προβλημάτων που μπορούν να προκύψουν στη διαδικασία τροφοδοσίας για τα τρόφιμα. Υπάρχουν και θέματα προστασίας ε, των φυσικών πόρων, τεχνολογία. Για όλα αυτά εξετάσαμε ποια είναι τα κύρια διεθνή ε, πρότυπα και τα συνοψίσαμε για να μπορούν να ληφθούν υπόψη στις πολιτικές των εταιριών για υπεύθυνη εταιρική στάση. Και επίσης υπάρχει ιδιαίτερο τμήμα για τη δέουσα επιμέλεια. Υπάρχουν πέντε βήματα. Βοηθάμε τις επιχειρήσεις λοιπόν να συμμορφωθούν με την ε, δέουσα επιμέλεια. Θέλουμε κατόπιν να υπάρξει ένα πιλωτικό πρόγραμμα με τις ενδιαφερόμενες εταιρείες και αυτό θα τις βοηθήσει να τηρήσουν την νομοθεσία και τα πρότυπα. Και θέλω να ασχοληθώ και με τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που συνδέεται και με τον προηγούμενο γύρο ομιλίων. Όπως διαπιστώσαμε, εάν δεν υπάρχουν επαρκή νομοθετήματα, Κάποιες επιχειρήσεις βέβαια μπορεί να κάνουν ακόμη και περισσότερα από ό,τι προβλέπει η νομοθεσία, αλλά για να τηρούν τι προδιαγραφές όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να υπάρχει ε, δεσμευτική νομοθεσία. Και ακόμη και αν είναι δεσμευτική μπορεί να είναι ευέλικτη η εφαρμογή της νομοθεσία Να μην γίνεται δηλαδή με λατρικό τρόπο. Και νομίζω ότι για παράδειγμα ο νόμος για τη σύγχρονη δουλεία δείχνει πώς μπορεί να γίνει αυτό. Ζητείτε από τις επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι έχουν κάνει την δέουσα επιμέλεια, αλλά το κάνουν με ανοιχτό τρόπο, ούτως ώστε και οι καταναλωτές να έχουν πληροφόρηση, ούτως ώστε όλοι να επιδιώκουν να έχουν τη βέλτιστη προσέγγιση, να είναι αγώνας προς τα πάνω. Έτσι οι επιχειρήσεις είναι πιο διαφανείς και οι καταναλωτές μπορούν να τις πιέσουν για να βελτιώσουν τις πρακτικές τους. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την άποψη του ΩΣΑ, τι κατευθυντήριες γραμμές και κάποιε συμβουλέ προ του νομοθέτε. Τι έχει όμω να πει η βιομηχανία. Με χαρά μου καλωσορίζω τη Βαλέρια Ραμικόνη, η οποία είναι συντονίστρια ε, για ευρωπαϊκά ε, ζητήματα από την Global Sea Alliance. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα. Θα σας κάνω μία σύντομη παρουσίαση και μία σύντομη εισαγωγή για το τι είναι το καριτέ και ποια είναι η αλυσίδα αξίας του και πώς ε, εργαζόμαστε στην Global Sea Alliance. Ο οργανισμός μας είναι ε, μία ένωση παραγωγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Προσπαθούμε να προωθήσουμε ε, κοινά πρότυπα και βιωσιμότητα στον ε, χώρο της καλλιτικής βιομηχανίας και της βιομηχανίας τροφίμων για το Καριτέ. Το 2011 συσταθήκαμε, τώρα έχουμε 390 μέλη από 30 χώρες στα μέλη μας ανήκουν διεθνείς επιχειρήσεις όπως το Body Shop, η Nestlé, διεθνείς και ε, τοπικές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, Ινστιτούτα και κοοπερατίβες αγροτικές. Επόμενη διαφάνεια. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι ακριβώς είναι το καριτέ, καλύτερα θα ήταν να σας έκανα μια περιγραφή των δύο κύριων χαρακτηριστικών αυτού του καρπού. Καταρχάς, το καριτέ καλλιεργείται μόνο σε μια περιοχή του κόσμου περίπου 2 δισεκατομμύρια δέντρα καριτέ φύονται ε, από μόνα του στην Δυτική και Κεντρική Αφρική. Από τη Σενεγάλη μέχρι το Νότιο Σουδάν είναι η ακτίνα του φυτού αυτού. Όπως είπα, τα δέντρα αυτά είναι αυτοφυή, δεν υπάρχουν φυτίες δηλαδή, δεν μπορούν να καλλιεργηθούν. Ε, υπάρχουν μαζί με άλλες καλλιέργειες στα αγροκτήματα. Τα δέντρα αυτά έχουν καρπούς, οι οποίοι μοιάζουν με μικρό μάγκο, έχουν σκληρό ε, φλοιό και μέσα πυρήνες. Οι πυρήνες μοιάζουν με μικρούς πυρήνες από ροδάκινα, οι οποίοι συλλέγονται, επεξεργάζονται, έτσι ώστε να ε, αποκομίσουν το λάδι, καριτέ. Και η διαδικασία αυτή συλλογή και επεξεργασία των επιρρήνων για το βούτυρο καριτέ γίνεται από γυναίκες. Οι γυναίκες λοιπόν βρίσκονται στην καρδιά της αλυσίδα αξίας του καριτέ. Περίπου 16 εκατομμύρια γυναίκες ασχολούνται με τη συγκομιδή αυτών των καρπών και είναι ένα βασικό ε, εισόδημα για τις οικογένειες ε, ορισμένων από τις φτωχότερες περιοχές της Αφρικής. Να σας δώσω τώρα μία εικόνα για την αλυσίδα αξίας του καριτέ. Στην κορυφή έχουμε τις γυναίκες. Μετά. Κάποια στατιστικά στοιχεία. Κάθε χρόνο έχουμε περίπου 1,2 εκατομμύρια πυρήνες ως παραγωγή. 90% αυτών χρησιμοποιείται ε, στη βιομηχανία τροφίμων, ως ε, συστατικό δηλαδή, και 10% στην καλλιτική βιομηχανία. Μετά, επόμενη διαφάνεια. Πώς λειτουργούμε. Η Global Sea Alliance εστιάζει σε τρεις δράσεις. Προώθηση του καριτέ, ευαισθητοποίηση για την αλυσίδα αξίας του, προώθηση της ποιότητας, δηλαδή δημιουργία προτύπων ποιότητας για τους πυρήνες και όλα τα προϊόντα που περιέχουν καριτέ και ε, διασφάλιση της βιωσιμότητας της αλυσίδας αξίας. Ε, αυτό μέσω μιας πολυμερούς προσέγγισης από ενδιαφερόμενους. Το 2011 λοιπόν άρχισε η διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος με κατευθυντήριες γραμμές και ε, που αφορά τη βιωσιμότητα. Και εμείς διευκολύναμε αυτή την ε, πολυμερή διαβούλευση. Αυτό επιθυμούσαμε. Συγκεντρώσαμε δηλαδή όλους τους ε, φορείς ε, που δραστηριοποιούνται με το καριτέ. Βλέπετε εδώ στα δεξιά τον εκπρόσωπο από την Hershey, την εταιρεία αυτή τροφίμων. Βλέπετε μία εκπρόσωπο από το Body Shop εκπρόσωπο από τοπική ΜΚΟ και στην ε, αριστερή άκρη με τα κίτρινα ε, μία εκπρόσωπο από μία οργάνωση γυναικών, η επικεφαλής μιας οργάνωσης γυναικών. Γίνεται λοιπόν αυτή η διαβούλευση και περίπου μετά από τρία χρόνια καταλήξαμε ε, σε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για τη βιωσιμότητα. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν τέσσερις κύριες προτεραιότητες. Χειραφέτηση των γυναικών, αξιοπρεπή συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και Τώρα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς στην αλυσίδα αξία του Καριτέ πρέπει να συνεργαστούν έτσι ώστε να ε, συμμορφωθούμε τις κατευθυντήριες γραμμές. Αυτό εδώ είναι ένα παράδειγμα από τις αξιοπρεπείς ε, συνθήκες εργασίας και τις αρχές που τις διέπουν. Τώρα, για να εφαρμόσουμε αυτό, αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές για την ε, βιωσιμότητα, εντοπίσαμε με όλους τους συνεργάτες μας περίπου έξι έργα τα οποία ε, μπορούμε να εκτελέσουμε. Τα λέμε αυτά work streams. Ε, εκπαιδευτική Εκπαίδευση και κατάρτιση στις επιχειρήσεις, ε, για τις γυναίκες, ε, πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και την υγεία, έργα ε, συντήρηση, διαχείριση των ε, φυτών καριτέ και έρευνα και ανάπτυξη αναπαραγωγικού υλικού. Για να μπορέσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε σωστά όλα αυτά τα προγράμματα, χρειαζόμαστε τη βοήθεια και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αυτή τη στιγμή οι ιδιωτικές επιχειρήσεις έχουν συνεργαστεί μαζί μας για την εφαρμογή αυτών των ε, work streams. Υποφάλουν εκθέσεις κάθε χρόνο στην ε, Global Sea Alliance σχετικά με την εφαρμογή και την εξέλιξη αυτών των προγραμμάτων, αλλά και με τις ε, κυβερνήσεις προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να, να δημιουργήσουμε συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να, να επιτύχουμε τους στόχους μας, δηλαδή να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες ζωής των γυναικών αυτών στην Ήπεθρο και να δημιουργήσουμε υψηλή ποιότητα πρότυπα για όλα τα προϊόντα που περιέχουν καριτέ προς ε, όφελος των καταναλωτών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ μου φαίνεται ένα πολύ καλό παράδειγμα. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πάντα. Είμαι σίγουρος όμως ότι ο Μάρκ Μέις τώρα θα μας αναφέρει τις αντίθετες περιπτώσεις. Είναι υπεύθυνο πολιτικής ε, μιας βελγικής μη κυβερνητικής οργάνωσης 11-11-11. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαι εδώ εκ μέρους της Concord, της Ευρωπαϊκής Ομοσπανδίας για του μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, που εκπροσωπεί 2.600 ΜΚΟ στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όντως είμαι υπεύθυνος για το εμπόριο στη βελγική πλατφόρμα, όμως μιλώ εδώ εκ μέρους της Concord και έχω λάβει πολλές πληροφορίες από τα μέλη πριν έρθω εδώ. Το ε, μήνυμα από τα μέλη της Concord είναι τριπλό. Πρώτον, η Concord ενδιαφέρεται πολύ για τους αγρότες που σε μικρή κλίμακα δραστηριοποιούνται και ζηλεύουν την αξία που δίνεται στις αλυσίδες αξίας. Αυτοί εκπροσωπούν το 60 με 70% των τροφίμων παγκοσμίω ε, που δεν διοχετεύονται στις παγκόσμιες αλυσίδες αλλά στις τοπικές. Ο ρόλος ε, των μικρών γεωργών ε, για την επίτευξη της Ατζέντα 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης είναι να έχουν μια βελτιωμένη παραγωγή ώστε να δώσουν στον κόσμο την τροφή που χρειάζεται αλλά και να βοηθήσουν τον κόσμο τον αναπτυσσόμενο να κάνει την απαραίτητη μετάβαση. Αυτό που ζητούμε από τους μικρούς γεωργούς λοιπόν είναι φυσικά από τη μία να έχουν υποστήριξη από τις ε, κυβερνήσεις τους αλλά και από τη διεθνή κοινότητα δωρητών και για την ε, πολιτική εμπορίου θέλουμε να εμπλέκει τους μικρούς γεωργούς εξ αρχής να έχουν μεγαλύτερο λόγο στην διαμόρφωση της πολιτικής εμπορίου πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις ε, και όταν γράφονται οι εντολές. Θέλουμε η πολιτική εμπορίου να διασφαλίζει ότι υπάρχει το δικαίωμα προστασίας των γεωργών και υποστήριξης αυτών, αλλά και να υπάρχει πρόσβαση στη γη και στους σπόρους. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον, μόνο 10 με 12% της γεωργικής παραγωγής ανά τον κόσμο καλύπτεται από τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας. Διεθνέ εμπόριο. Αυτές οι αλυσίδε κυρίω ξεκινάνε από εμά, από τι δικέ μας ανάγκες και τα πράγματα που εμείς θέλουμε. Τις πρώτες ύλε που ζητούμε, τα βιοκαύσιμα, τα τρόφιμα, τον καφέ, τις καρύδες, ε, το... οτιδήποτε. Θα πρέπει λοιπόν να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το αποτύπωμά μας. Πολλές χώρες όπως η Ολλανδία καταναλώνουν τρεις φορές παραπάνω από ό,τι οι ίδιες παράγουν. Έτσι ζητούν να εισάγουν και πιέζουν ευάλωτες περιοχές και οικοσυστήματα, ε, ειδικά μικρούς αγρότες. Αν θέλουμε λοιπόν να μιλάμε για βιώσιμες αλυσίδες αξίας, θα πρέπει να μιλάμε για ίδια κατανάλωση των, της δικής μας παραγωγής. Δεύτερον, για το πώς θα γίνουν πώς πιο βιώσιμες οι αλυσίδες. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να γίνει αυτό, διότι υπάρχουν ε, περιβαλλοντικά προβλήματα λόγω των φυτιών, οι γεωργοί παίρνουν χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους, εκμετάλλευση των εργαζομένων στις φυτίες. Αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχουν διάφορα μέσα για να επιτύχουμε πιο βιώσιμες αλυσίδες. Υπάρχει μεγάλη εθελοντική ε, δουλειά που γίνονται. Πολλά από τα μέλη μας ε, το κάνουν αυτό. Υπάρχει ένα κίνημα που ήταν πρωτοπόρο για τη δημιουργία σταθερών τιμών στην παγκόσμια αγορά, ή το κίνημα Φρέντρικ, το οποίο προσπαθεί να φέρει ε, τη βελτίωση από το επίπεδο των γεωργών μέχρι και τα σούπερ μάρκετ. Θέλουμε λοιπόν μέσα από τα ετικέτες Fair Trade δίκαιο εμπόριο να πετύχουμε αυτούς τους στόχους, γιατί πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια. Ε, πολλοί λοιπόν ε, εκπρόσωποι του Fair Trade έχουν ε, ασχοληθεί με διάφορες βιομηχανίες και έχουν μιλήσει για το θέμα της παιδικής εργασίας. Έχουμε την Διεθνή Οργάνωση για που ασχολείται με αυτό. Έχουμε επίσης ε, και τα βελγικά σούπερ μάρκετ που έχουν άμεση επαφή με τους παραγωγούς και δίνουν τα μέσα για τη βελτίωση της βιώσιμης παραγωγής από τους μικρούς γεωργούς. Η ίδια η βιομηχανία λοιπόν έχει εισαγάγει τις δικές της ετικέτες. Υπάρχουν ε, εταιρείες ε, που εμπορεύονται μπανάνες και έχουν βάλει την ετικέτα τους σε φυτίες, διεθνείς οργανισμοί, ο ΣΑ για παράδειγμα, που δίνουν τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες για τις εταιρείε. Όμως, μέχρι εδώ μπορούν να φτάσουν τα εθελοντικά προγράμματα. Θέλουμε περισσότερη λοιπόν επιβολή της εφαρμογής καλών πρακτικών επιχειρηματικών προοπτικών. Τι πρέπει να γίνει. Καταρχάς να υπάρχει μεγαλύτερη πίεση στις κυβερνήσεις, να υπάρχει το κεφάλαιο της διώσιμης ανάπτυξης σε όλες τις συμφωνίες εμπορίου και να είναι και εφαρμόσιμο και να εκτελείται. Επίσης να αντιμετωπίσουμε τις χειρότερες μορφές κατάχρησης όπως την παιδική εργασία, την άρνηση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Υπάρχει επίσης το πρόβλημα που είδαμε στο παρελθόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συνάψει συμφωνίες με χώρες που παραβιάζουν τα ανθρώπινα και τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά οι συμφωνίες να γίνονται. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες να ασκηθεί η πίεση στις κυβερνήσεις αυτές πριν τη σύναψη της συμφωνίας. Ας πούμε, στην Κολομβία και στο Περού υπήρχε ένας οδικός χάρτης που ζητήθηκε να εφαρμοστεί από τις χώρες αυτές ε, ε, ήταν πολύ πιο λεπτομερής από ό,τι ήταν συνήθως και ίσως το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και με άλλες χώρες. Υπάρχει τώρα αυτό το βιβλίο του Oliver de για την βιώσιμη ανάπτυξη, δεν ξέρω αν το ξέρετε, εξηγεί ότι ακόμα και με τους κανόνες του ΠΟΕ μπορεί κανείς να πάρει μονομερή μέτρα ώστε να βοηθήσει στο βιώσιμο εμπόριο με βάση τα διεθνή στάνταρα, αν υπάρχει μια μεταβατική περίοδος, αν υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες που εμπλέκονται και αν τα έσοδα που δημιουργούνται μας βοηθούν να ε, επιτύχουμε τους στόχους. Αυτά πρέπει η Ευρώπη να τα διερευνήσει για να μπορέσει να τηρήσει και τα κοινωνικά και τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Υπάρχει εδώ αυτό το βιβλίο και πρέπει να το δείτε. Δεύτερον, τα περισσότερα από τα μέτρα ε, ναι μεν ε, λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις, αλλά χρειάζεται και μεγαλύτερη πίεση στις εταιρείες. Αν μιλάμε για το παράνομο λόμπινγκ, ε, ε, συγγνώμη, την παράνομη ξύλευση και άλλα τέτοια παράνομα προϊόντα στον κόσμο όπως ε, μπανάνες ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να μην εμπορευόμαστε με παράνομες τέτοιες φυτίες και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ πολύ. Ανελίτς, μία πρώτη σύντομη ερώτηση. Ανελίτς. Και εγώ μόνο ένα λεπτό θα χρειαστώ η Επιτροπή προσπαθεί να στηρίξει ορισμένες αφρικανικές χώρες για να επενδύσουν. Ερώτηση. Το προβλέπετε αυτό. Θέλουν να υπάρξουν περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις Το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι η Επιτροπή θέλει να ενθαρρύνει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Και τι θεωρείτε ότι θα επιτύχει. Θεωρείτε ότι η πρόθεση της Επιτροπής να δεσμευθούν τα κράτη-μέλη ότι θα κάνουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις έχει έννοια, θα αποδώσει, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα επιχειρήσω να είμαι σύντομο γιατί πρέπει να φύγουμε για για τον τριμερή διάλογο για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων. επίκειται το επόμενο G20 στο Χαντζού και οι αλυσίδες αξίας ε, είναι ένα από τα βασικά θέματα που θα ζητηθούν. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να κάνει το G20 για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες σας, αυτά που μόλις συζητήσαμε. Θεωρείτε ότι το G20 μπορεί να συμβάλλει στην επίλυσή τους σε διάφορους τομείς και εκεί που δεν έχουμε επαρκή ρύθμιση. Ο πρόεδρος. Έχουμε πολλές ε, γεωργικές εισαγωγές από τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, περίπου 70%. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ΑΕΠ τους ιδιαίτερα στη Δυτική Αφρική. Κάποιες χώρες έχουν ΑΕΠ ε, έως και 80% από τις εξαγωγές τους προς την Ένωση. Αλλά βέβαια το νομίσμα έχει δύο όψεις. Ε, απ' τη μια είναι οικονομικά σημαντικό για τις χώρες αυτές να συνεχιστούν αυτές οι εισαγωγές, αλλά πρέπει να είναι και βιώσιμες. Πώς μπορούμε να αντιστρέψουμε την αλυσίδα για να ωφελούνται επαρκώς. Να μην διατηρείται μόνο το ΑΕΠ, αλλά να υπάρχει ανάπτυξη. Λοιπόν, τώρα να απαντήσουμε αντίστροφα. Πρώτος ο Μάρκ. Δεν ξέρω αυτή την πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη προηγούμενη εβδομάδα στην οποία αναφερθήκατε. Λυπάμαι. Θα το κοιτάξουμε ω οργάνωση Concord και θα τοποθετηθούμε για τι ε, λιγότερο αμπτυγμένε χώρε και τα προϊόντα του. και το πώς μπορούμε να το συνδυάσουμε με την βιώσιμη ανάπτυξή τους. Ε, δύσκολο θέμα. πολλές από τις αγωγές είναι κακάο και καφές. Και αυτά κυρίως παράγονται από μικρές εκμεταλλεύσεις. Και οι μικρές εκμεταλλεύσεις χρειάζονται πολύ περισσότερη στήριξη για να μπορούν να εμπορευτούν τα προϊόντα τους. Ε, κάποτε στη Δυτική Αφρική όλη η αλυσίδα του κακάο οργανωνόταν από, την, ε, από τις κυβερνήσεις. Έδιναν τα ζυζανιοκτώνα, έδιναν όλο τον εξοπλισμό, είχαν τις αποθήκες αλλά έγιναν ε, πολιτικές ε, διαθροτικών προσαρμογών και τώρα ναι μεν ε, έχουν μεγαλύτερο ποσοστό στην παγκόσμια αγορά αλλά έχει αυξηθεί και το κόστος παραγωγής. Κάτι πρέπει να γίνει λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να υπάρξουν ελάχιστες τιμές. Υπάρχουν γενικώ, αλλά είναι ενδεικτικές. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι γεωργοί θα λαμβάνουν μια σωστή τιμή για να μπορούν και να επενδύσουν περισσότερο. Και δεν θα χρειαστεί να υπάρχει παιδική εργασία και άλλες ε, απαράδεκτες μορφές ε, εργασίας. Όπου στην αρχή της αλυσίδας είναι οι μικρές εκμεταλλεύσεις, αυτή την προσέγγιση χρειαζόμαστε. Αν ασχολείστε τώρα με μεγάλες φοιτίες, είναι άλλο το θέμα, όπως είπε και ο Γιώργος. Τα συνδικάτα πρέπει να μας ενημερώνουν για το τι συμβαίνει. Πρέπει να τα αυτιά και τα μάτια μας. Πρέπει να βοηθήσουμε τα συνδικάτα να έχουν περισσότερες δυνατότητες, να μας δώσουν αυτή την ενημέρωση και να πιέσουμε και τις κυβερνήσεις για να ε, γίνονται σεβαστές οι κοινωνικές προδιαγραφές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Βαλερή. Σας ευχαριστώ. Ναι, γνωρίζουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις πρωτοβουλίες μάλλον, που θα ενισχύσουν την συμβολή του, δημόσιου, του ιδιωτικού τομέα. Και συμφωνούμε. Διότι και εμεί αναπτύσσουμε τέτοιες δράσεις από το 2011. Για μας, για την αλυσίδα αξίας του Καριτέ, βλέπουμε ότι έχει αποτέλεσμα αυτό. είναι πάρα πολύ σημαντικό το ε, του Καριτέ, διότι περίπου το, 12% του εισοδήματος ε, των οικοκυριών αυτών προέρχεται από αυτό. Δεν αρκεί όμως. Χρειάζεται βελτίωση αυτού του ποσοστού όχι μόνο επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες διαβίωσης των γυναικών εκεί, όχι μόνο για τη βιωσιμότητα, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και την ε, βιομηχανία. Διότι εάν η βιομηχανία διαπιστώσει ότι το καριτέ δεν ε, αποφέρει κέρδος, τότε θα τα κόψουν τα δέντρα. Θα τα κόψουν διότι θα υπάρχουν άλλα πιο κερδοφόρα ε, φυτά υλικά ή η ξυλία τους θα είναι πιο πολύτιμη από τον καρπό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά, όχι μόνο για την ε, διασφάλιση της βιωσιμότητας, αλλά και για την ε, δέσμευση της ε, βιομηχανίας για την βελτίωση των συνθήκων. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι η συνεισφορές αυτές έχουν αυξήσει τα κέρδη των γυναικών κατά 51% για κάθε σακούλα από πυρήνες καλύτερα. Είναι λοιπόν μια τεράστια βελτίωση αυτή, διότι τα χρήματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αγοράσουν τρόφιμα, για να πληρώσουν δίδακτρα για τα παιδιά τους και ούτω καθεξής. Η συνεισφορά λοιπόν του ιδιωτικού τομέα είναι ευπρόσδεκτη και φυσικά και συνεισφέρει στην αλυσίδα αξίας και στην βιωσιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Καρολίν Νταβίδ. Ναι, θα απαντήσω σε δύο ερωτήσει. Στην πρώτη για του ε, G20 και στην δεύτερη ανάμεσα στις ε, συναλλαγέ ανάμεσα στην ε, ΔΕΛΤΑ ανάπτυξη και τις επιχειρήσεις. Τώρα, G20. Συμμετείχαμε σε όλες τις διαπραγματεύσει. Δεν έχουμε όμως και πολλές ελπίδες για το για να μπει ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων η βιωσιμότητα. Την επόμενη φορά θα προεδρεύσει η Γερμανία στο G20. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει, ε, υπάρχει μια ελπίδα να μπει το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Τώρα, αυτές οι σχέσεις ανάμεσα στις, ε, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, να σας πω ότι έχουμε διαπιστώσει μετά από μελέτες ότι τουλάχιστον σε επίπεδο επιχειρήσεων μπορούν με, να υποφεληθούμε από τις πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Μία πρόσφατη μελέτη που αφορούσε περίπου 10.000 γαλλικές εταιρείε έδειξε ότι υπήρχε μία διαφορά 13% ανάμεσα σε εταιρείε που ακολουθούσαν καλές πρακτικές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και σε εκείνες που δεν ακολουθούσαν τέτοιες πρακτικές. Υπάρχει λοιπόν μια αισθητή διαφορά και αυτό φαίνεται και από τις έρευνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Σάντρα, άκουσες τους πάντες. Έμαθε κάτι καινούριο, έχεις κάποιες καινούργιε σκέψει. Ναι. Και ευχαριστώ όλους γι' αυτό. Θα ήθελα όμως να επιστρέψω σε κάτι το οποίο ε, ακούστηκε εδώ, την πολιτική θέληση. Λοιπόν, τι μπορεί καταρχάς να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρωτοβουλία, όπως είπαμε. Πηγαίνετε πίσω στις πατρίδες σας, μιλήστε, ενημερώστε. Αυτό είναι πολιτική θέληση κατά έναν τρόπο. Τώρα, ε, οι κυβερνήσεις, παρότι πολλές φορές μπορεί να έχουν πολιτική θέληση, τους λείπει η δυνατότητα ανάπτυξης και πολλές φορές έχουν και κάποια θεματάκια και με τι εργασιακέ συνθήκε, αλλά και με την Ευρώπη. Ε, τώρα, να σας μιλήσω για το 50 for Freedom. Είναι κάτι που αφορά περισσότερο τη διακίνηση ανθρώπων, αλλά έχει σχέση και με αυτά που συζητάμε. Ας μην νομίζουμε ότι είμαστε τόσο τέλειοι και ότι μπορούμε να γυρίζουμε τον κόσμο κηρύσσοντα το σωστό. Εάν η G20 αποδεχθεί αυτές τις, ε, αυτά, τα, αυτά τα αιτήματα, τότε θα αναγκάσει και την Κίνα να τα δεχτεί. Σήμερα το απόγευμα έμαθα κάτι το οποίο ήδη γνώριζα. Βλέπω ότι πολλές φορές συγχέουμε διαφορετικά πράγματα. Και επιτρέψτε μου μία περισσότερο πολιτι... Ε, προσωπική παρά πολιτική δήλωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μιλάμε τώρα για εργασιακά πρότυπα. Υπάρχουν όμως υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας. Δεν έχουν καμία σχέση με την ε, κοινωνική εταιρική ευθύνη. Τι είναι η εταιρική κοινωνική ευθύνη, αυτό που συζητούσαμε και με τον Νίκο. Ας πούμε, μία εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί ένα κυκλωμένο χαρτί αυτό είναι κάτι εθελοντικό και σίγουρα ο εθελοντικός χαρακτήρας είναι προτιμότερος και έχει καλύτερα αποτελέσματα. Δεν είναι όμως κατά ανάγκη αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να ε, έχουμε μία βιώσιμη αλυσίδα αξίας. Ε, τι άλλο, έλεγχος, ποιος ελέγχει για το αν εφαρμόζονται αυτά τα πρότυπα. Ζητώ συγγνώμη εάν το σχόλιο μου είναι πιο προσωπικό, και δεν μιλώ τόσο με την ιδιότητα της ε, εκπροσώπου της Επιτροπής, όμως βλέπω ότι υπάρχουν όντω διαφορές ανάμεσα στον τομέα της ένδυσης και στον τομέα της ε, γεωργίας. Υπάρχουν άλλες δομές. Ε, στην περίπτωση της γεωργίας υπάρχουν γυναίκες που θρέφουν οικογένειες. Θα μου πείτε και στην περίπτωση της Ραναπλάζα είχαμε γυναίκες. Αλλά αυτό είναι πιο πολύ θέμα συνδικαλιστικό. Γι' αυτό λοιπόν σας είπα ότι το θέμα της ασφάλειας, το ε, εξετάσαμε, αλλά υπάρχουν ακόμα ελλείψεις. Σήμερα το απόγευμα, προσωπικά, βρήκα στοιχεία τα οποία ε, αποτελούν μια πάρα πολύ καλή αφετηρία για περαιτέρω συζητήσεις και νομίζω πως έχει παίξει ρόλο και η Ολλανδική Προεδρία σε αυτό, διότι η καινοτόμως πρωτοβουλία τους βοήθησε πολύ. Ένας ε, υπουργός ανέλαβε και θέματα εμπορίου και θέματα ανάπτυξης. Συνδέθηκε δηλαδή αναπτυξιακή συνεργασία με το εμπόριο, το οποίο είναι πιστεύω πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν που έμαθα και αποκόμισα αυτό το απόγευμα είναι ότι όλοι θα γυρίσετε στα σπίτια σας έχοντας διδαχθεί κάτι και πρέπει να κοιτάζουμε όχι μόνο τι κάνουν οι άλλοι αλλά τι κάνουμε και εμείς. Ευχαριστώ. Όντως, το θέμα της συνέχειας είναι κεντρική σημασίας και ο έλεγχος, η παρακολούθηση επίσης. Αλλά επί της αρχής να πω ότι είμαι πλήρως πεπισμένος ότι το να επικεντρωθούμε στις παγκόσμιες αλυσίδες ε, αξίας ε, θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι για τη μελλοντική πολιτική εμπορίου. Αν βρούμε σήμερα ένα συμβασμό για τα μεταλλεύματα από τις τα χώρες όπου υπάρχουν σειράξεις και γενικά τέτοιες πρωτοβουλίες, θα έχουμε και άλλες ε, πρωτοβουλίες όπως για την ξυλία, έχουμε την ένδυση και θα προωθήσουμε εκεί για κάποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες. Θα είμαστε πάντοτε λοιπόν στο πλευρό σας για να μπορέσει να γίνει σωστή μεταχείριση των παγκοσμίων αλυσίδων αξίας που θα συμφέρει τους ντόπιου παραγωγούς και αυτό θα είναι και ο στόχος της πολιτικής εμπορία που θα βασίζεται στην αξία. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους εμπειρογνώμονες διότι ε, συνέβαλαν ιδιαίτερα στην επικοδομητική αυτή συζήτηση ένα χειροκρότημα. Θα δώσουμε τις ομιλίες, τις παρουσιάσεις στα μέλη και θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τα μέλη της Επιτροπής αύριο το πρωί στις 9 και πάλι εδώ.